Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Καλημέρα κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε πολλούς συνάδελφους ήδη εδώ, μπορεί να μην έχουμε ολομέλεια. Αλλά νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι εδώ για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Όπως ε, γνωρίζετε πάντοτε στις ψηφοφορίες χρειαζόμαστε και την ε, κάρτα μας για να ψηφίσουμε. Και εγώ χρειάζομαι τη δικιά μου. Ξεχάσατε την κάρτα, ε, θα είναι δύσκολο άμα την έχει ξεχάσει. Εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε πιο πολύ μαζί μας την κάρτα μας, Dann kommen. Ας ε, περάσουμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία για την έκθεση του Άλλος Πέτρελε σε ό,τι αφορά την έκθεση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρτίνου Ευρωπαϊκή Σύμπραξη. Έχουμε τον κατάλογο ψηφοφορίας που ξεκινάει με την τροπολογία 31, η οποία είναι ταυτόσιμη με την τροπολογία 32. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρινέται. 33 και 34 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 α, καταπίπτει 37 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 38 και 42. Ταυτόσημες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή μετά περνάμε στην 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50. Θέλει να πει κάτι ο συγητή σε σχέση με την 50. Αν ο συγητή είναι υπέρ, μπορώ να σα το πω εγώ, όχι λοιπόν κατά, είναι υπέρ. Ε, στην τροπολογία Σεντερλάνια. Άρα λοιπόν ψήφι υπέρ για τροπολογία 50. Κατά, άποχες, εκρίνεται. 51. Με oral amendment, προορική τροπολογία από τον εισηγητή. Ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 9 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή Τώρα, συμβασμός, συμβαστική τροπολογία, υπαριθμόν 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μενάμε τώρα στη 56, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57, με την τροπολογία του εισηγητή, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 58 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. 59 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτή. 60 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. μετά από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα της γυναίκα μια τροπολογία με split vote εδώ ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ για το πρώτο τμήμα της τροπολογία, ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται τρίτο τμήμα καταπίπτει συμβαστική τροπολογία 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 4 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 5 ψήφι υπέρ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 ψήφι υπέρ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 απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θεμ 8 κλιματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 74 με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 15 καταπίπτει, οπότε περνάμε στην 75. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 17 με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 3 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατά καταπίπτει περνάμε τώρα στην τροπολογία 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φεμ α ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, κυρία μα βλέπετε, έχουν εγκριθεί πολλές τροπολογίες. Όλα καλά πάνε για σας. Ήτρε Β. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φεμ Δ. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επιτροπή Διοικών Ε ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή Γυναικών F. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά περνάμε στην τροπολογία 10 και 11 που είναι ταυτόσιμες με τμηματική ψηφοφορία από S&D ε, πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 και η Επιτροπή Γενικών J είναι ταυτόσιμες. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 16 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 17 και η Επιτροπή Γενικών G είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται και αυτές. 18 και Επιτροπή Γυναικών ΚΑΠΑ ταυτόσιμες ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 19 και Επιτροπή Γυναικών ΕΛ είναι ταυτόσιμες ψήφι Κατά. Αποχές. Και αυτή απορρίπτεται. Επιτροπή Γυναικών μη ψήφι Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπή εν ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 22 και 23 είναι ταυτόσιμε. ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρινόνται Επιτροπή Γυναικών ΆΗ ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 και 25 ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 26 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 27 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Περνάμε τώρα λοιπόν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της χθε Έναρξη λοιπόν τη ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. 56 λοιπόν ψήφοι υπέρ, 56 ψήφισαν, καμία αρνητική ψήφος και καμία αποχή. Τα ζητημά μας συγχαρητήρια λοιπόν στον συνάδελφο Πέτερλε και τις ευχές μας για κάθε επιτυχία στην καταπολέμηση του καρδίνου, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και έξω από αυτήν. Ε, γνωρίζω πόσο δραστήριος είναι όλος Πέτρελε σε αυτόν τον τομέα. Και τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσους συνεργάστηκαν για αυτήν την έκθεση και την γραμματεία. Περνάμε λοιπόν τώρα από τον καρκίνο στη Βαλτική θάλασσα και η συγκίτρια θα ήθελε να πει κάτι. Παρακαλώ, Άννα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, σίγουρα άφησα κατά μέρος κάποιες τροπολογίες. Να εξηγήσω γιατί. Στην τροπολογία 2 ξεκινάμε. Θα ήθελα στην τελευταία πρόταση να αφήσουμε ένα είδος ε, ψαριού. Τις δύο τελευταίες λέξεις. Θα ήθελα να αφήσουμε λοιπόν τις δύο τελευταίες λέξεις. Το σίκο του Ατλαντικού Μπακαλιαράκη. Γιατί, κατά τα άλλα είμαι ικανοποιημένη με την τροπολογία. Καταρχάς ε, προβληματίστηκα για το κατά πόσο θα πρέπει να μείνει η Ρωσία, να αναφέρεται η Ρωσία. Αλλά σε τελική ανάλυση συμφωνώ με την ε, τροπολογία αυτή. Στο 16 τώρα. Μιλάμε για τα καθαριστικά. Με την προφορική τροπολογία αυτή συμφωνώ. Και τέλος έχουμε την τροπολογία 10 η οποία είναι ανοιχτή. 18, συγγνώμη. Μία μικρή προσθέκη. Υπάρχει μία αρχή του ρηπαίνων πληρώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο, ο πιο μεγάλος ρηπαίνων στην Βαλτική είναι η Ρωσία. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε μία μικρή προσθήκη στο σημείο αυτό στην τροπολογία 18. Αν θα μπορούσαμε να βρούμε μια τέτοια προσθήκη για να αναφερθεί το ρηπαίνον πληρώνει και να συμπεριληφθεί και η Ρωσία. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να πω. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος. Λέει ο Πρόεδρος, όμως με αυτή την προσθήκη, αυτή τη γενική, δεν μπορούμε να περάσουμε σε ψηφοφορία. Θέλουμε συγκεκριμένη προφορική τροπολογία, αλλά μάλλον δεν υπάρχει αυτή. Καλή σκέψη, αλλά δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις σας. Μια διαγραφή από την τροπολογία 2 το συγκεκριμένο είδος που προτείνονται. Γιατί περιλαμβάνονται και άλλα ψάρια πέρα του γάδου. Να ψηφίσουμε λοιπόν τη 2 υπέρ. Κατά.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 Αποχές απορρίπτεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 16 με προφορική τροπολογία. Συγγνώμη, 15, διορθώνει η πρόεδρος, Γιατί 15, υπέρ. Γιατί 15 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Να το ελέγξουμε. Γιατί 15 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται λοιπόν η 16 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή να ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία έναρξη. Und geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. Σαφές το αποτέλεσμα. 54 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια για την εισηγήτρια που μένει πάνω στη Βαλτική και θα φροντίσει για την καθαρότητα της Βαλτικής. Να παραμείνει καθαρή η Βαλτική. Και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία, στο 11 της ημερήσιας διάταξης, το πρόγραμμα COSLO-DUI. Η Αντώνια Παρβάνοβα είναι η συγγήτρια. Καλημέρα. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόντες εισηγητές για τη βοήθειά τους. Είναι η πρώτη έκθεση που ανέλαβα ως εισηγήτρια. Θα ήθελα να φτάσω τον κύριο Πέτερλε. Μάλλον θα μου παραμείνει η... ο ειλικρινής θαυμασμός προς το τομό του. Να ευχαριστήσω και τους πράσινους για την υποστήριξή τους. Υπάρχουν κάποια σημεία διαφωνίας για τα 20 εκατομμύρια ευρώ για την ε, τελική απόρριψη των αποβλήτων. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε πλήρη συμφωνία. Ελπίζω μετά την ψηφοφορία να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Ωστόσο, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κυρία Παραβάνοβα. Ξέρετε, τα πράγματα τελικά κρίνονται πάντα στην ψηφοφορία. Θα διασπιστώσουμε λοιπόν τι θα επικρατήσει. Να ψηφίσουμε λοιπόν τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 11. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 35 υπέρ. Α, συγγνώμη πίπτη, Περνάμε στη 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. γίνεται μια πολύ ωραία και μάλλον ζωντανή συζήτηση στα τελικά, η οποία φαίνεται σας έχει προωθήσει. 13 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Η 38 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Η 14 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να το ελέγξουμε για την 40 παρακαλώ ένα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Schlossen. Πέρας. Ναι, Σωστό ήταν το αποτέλεσμα, οριακό μεν, αλλά σωστό. Εγκρίνεται. Η 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 42 καταπίπτει και αυτή και η 15 καταπίπτει, άρα η 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Οι δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. οι 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. περνάμε τώρα στην τέσσερα Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 22. Υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. Η 5 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Η 23 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Η 27 μετά, για το υπόλοιπο κείμενο, υπέρ λοιπόν για το υπόλοιπο κείμενο, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ. Αναφέρεται στην επόμενη σελίδα την καταπίπτη λοιπόν 28 και περνάμε στην 25 για το υπόλοιπο κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καταπίπτει 26. Στην 6 λοιπόν περνάμε υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Οι 29 και οι 30 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 31. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 8. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται και αυτή. Η 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Und ist geschlossen πέρασε. Συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια λοιπόν προ την εισηγήτρια. 47 η ψήφοι υπέρ, 7 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια για την έκθεση αυτή για το πρόγραμμα Κοζλοντουή, τους τον πυρηνικό σταθμό. Ήταν ένα δύσκολο κεφάλαιο. So. Wir sind bei dem Tagesordnungspunkt 12. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 12 της ημέρας σας διάταξης. Νέα τρόφιμα. Η συγκεκριμένη κατοίκα Λεωτάρ. Εξετάζουμε λοιπόν εδώ ένα σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια, την Δελιοτάτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα στην ε, συζήτηση δεν θα θέλω να σας δυσκολέψω. Στην πρώτη ανάγνωση η έκθεσή μου πέρασε στην Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία μόνο 15 ψήφοι Και γι' αυτό λοιπόν στη δεύτερη ανάγνωση αποφάσισα το κείμενο να παραμείνει όσο πιο κοντά γίνεται ε, στην έκδοση εκείνη, στο κείμενο εκείνο που είχε ψηφιστεί. Η οδηγία έχει ως σκοπό να ρυθμίσει την εισαγωγή νέων τροφίμων ε, στην αγορά για να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία της υγείας των ανθρώπων, αλλά και φυσικά να προστατευθούν η υγεία των ζώων, το περιβάλλον και τα συμφέροντα του καταναλωτή. Πρόκειται για νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν εφαρμόζονταν πριν από το 1990, για παράδειγμα 1997, για παράδειγμα εμ, νανοτεχνολογία, νανοηλικό. Χρειάζεται λοιπόν απαραίτητα επιστημονικός έλεγχος σε ό,τι αφορά αυτές τις νέες τεχνολογίες. Συμπεριλαμβάνονται οι τρόποι ελέγχου σύμφωνα με την ΕΦΣΑ και πριν ε, συμπεριληφθεί στον κατάλογο αυτό ένα τρόφιμο θα πρέπει να έχει περάσει από τον έλεγχο αυτό. Αν χρησιμοποιείται λοιπόν νανοτεχνολογίες για την παραγωγή ενός τρόφιμου θα πρέπει πρώτα να περνάνε από έγκριση τα προϊόντα αυτά. Το Κοινοβούλιο και σε προηγούμενα ψηφίσματα αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα που προέρχονται από το κρέας κλωνοποιημένων ζώων, γιατί προκύπτουν πάρα πολλά διλήμματα από την κλωνοποίηση ζώων σε ό,τι αφορά την ε, ζωή, την υγεία, την ευημερία των ζώων ανακύπτουν διοντολογικά προβλήματα και το Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί τότε ότι δεν έχει συζητηθεί αυτό επαρκώς ε, σε δημόσιες συζητήσεις και γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο τότε είχε αποφανθεί ότι θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή ρύθμιση σε ό,τι αφορά το κρέας αυτό των κλωνοποιημένων ζώων. Δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβανθεί στον, ε, κανόνα, στον κανονισμό αυτό για τα νέα τρόφιμα σε ό,τι αφορά τη διάθεση στην ε, αγορά δηλαδή του κρέατος αυτού. Και θεωρούμε ότι χρειάζεται πραγματικά μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό προτού αποφανθούμε. Το Συμβούλιο στην κοινή θέση του συμφωνεί και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του Κοινοβουλίου σε πολλά θέματα. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον ορισμό της νανοτεχνολογίας θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, αλλά και σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα, μόνο σε ό,τι αφορά την κλωνοποίηση. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε καταλήξει σε συμβιβασμό ακόμα, κοιτώντα την κοινή θέση του Συμβουλίου και την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια αποδεκτή λύση προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί ζητήσαμε και από τον νέο Επίτροπο να υποβάλει σύντομα μια νέα πρόταση για τη νέα νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα κλωνοποιημένα ζώα και απάντησε θετικά. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ε, πότε προβλέπετε να υποβάλλετε σχετική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ανοηλικά και την ανατεχνολογία. Συμφωνεί σε γενικέ γραμμέ το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο. Στην πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο σχετικό ορισμό, αλλά επειδή η νανοτεχνολογία είναι μια αγοργά αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη επιστήμη, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον να προσαρμόζεται αυτός ο ορισμός ανάλογα με τις εξελίξεις. στη ετικέτα των τροφίμων θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι πρόκειται για νέα τρόφιμα. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για τρόφιμα που έχουν ε, τύχη επεξεργασίας με ένα υλικό. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ε, στην ετικέτα. Για τα παραδοσιακά τρόφιμα, φρούτα, για παράδειγμα, ή για παραδοσιακά τρόφιμα φυσικής προέλευσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία απλοποιημένη για τα τρόφιμα αυτά. Θα ήθελα να ικανοποιηθεί και η αξίωση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις δοκιμές για τα ζώα, σε ζώα. Δοκιμές οι οποίε θα πρέπει να γίνονται όπω έχει υποστηρίξει το Κοινοβούλιο και στο παρελθόν, μόνο όταν δεν υπάρχει εναλλακτική άλλη λύση. Κατά τα άλλα, λοιπόν, ε, πιστεύω ότι αυτό θα τα πιο σημαντικά ε, ζητήματα τα οποία καλούμαστε να συζητήσουμε και ελπίζω γρήγορα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank an die Berichterstatterin. Ευχαριστούμε την ε, εισηγήτρια για την εισαγωγή που μας έκανε σε αυτό το ευρύ θέμα. Πρόταση λοιπόν για εξαίρεση ε, του κλωνοποιημένου κρέατος από το περιεχόμενο, αλλά ε, τα ζητήματα νάνο τεχνολογίας να τύχθουν μέσα. Στη σύσταση περνάμε ε, στην πρώτη στιγμή της ηγήτρας, την κυρία Πιλά Αγιούζου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία είναι πολύ σημαντική, σημαντική για την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και πολύ σημαντική για την μηχανία τροφίμων και δι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν ε, τα δύο σημαντικά ζητήματα όπως είναι τα νάνο υλικά, θα πρέπει να το μελετήσουμε το ζήτημα περαιτέρω δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε αυτά τα υλικά αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποια επιστημονικά επιχείρηματα για να το πετύχουμε. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι περισσότερο ιδεολογικού χαρακτήρα, το ζήτημα της κλωνοποίησης ε, των ζώων. Στα, τα, στα φυτικά, φυτικές ποικιλίες ε, φυτοορμόνες ε, ε, και κλωνοποίηση από εδώ και 25 χρόνια. αλλά και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα τώρα. Το ζήτημα της κλωνοποίησης ζώων σύμφωνα με την υπηρεσία ε, ασφάλειας τροφίμων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το μοναδικό ζήτημα εδώ είναι ηθικό ζήτημα, δεοντολογικό κλπ. Τώρα, Η πρώτη κλωνοποίηση είναι αυτή που δημιουργεί κάποια προβλήματα στα ζώα, αλλά μετά η κατάσταση ρυθμίζεται και δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος ανησυχίας. Μπορούμε, θα μπορούσαμε να το απαγορεύσουμε την κλωνοποίηση, αλλά αν υπάρξει απόρριση ο πλευρά του Κοινοβουλίου, όπως πρότεινε και ο Επίτροπος, είναι να κάνουμε μια ξεχωριστή πρόταση. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, επηρεάσουμε την νομοθεσία την οποία απαιτεί η βιομηχανία τροφίμων. Εντάξει, τώρα η κλωνοποίηση είναι μια νέα τεχνολογία, όπως ε, και παλιά προ 25 ετίας είχαμε την ε, κλωνοποίηση των φυτών, φυτικών ποικιλιών. Τώρα στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται ελάχιστα αλλά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στο μέλλον αυτή η τεχνική να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, διότι είναι μια τεχνική που βελτιώνεται και πως ε, βελτιώνεται και η ευημερία των ζώων. Αυτό επίσης που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να απαγορεύσουμε κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε στο μέλλον και δεν θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε σε τρίτες χώρες να μας προμηθεύουν με προϊόντα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, διότι πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε, να τα ανοιχνεύσουμε και δεύτερον, και, αυτό το λέω διότι δεν υπάρχει η χνηλεσιμότητα που υπάρχει στην Ευρώπη. Και ε, τέλος, εγώ θα απαγόρευα την πρώτη γενιά κλωνοποιημένων ζώων, αλλά όχι τους απογόνους. Και να πω και κάτι με το οποίο δεν συμφώνησα με τον Επίτροπο στην ακρόασή του, ότι θα πρέπει να γίνει μια χωριστή πρόταση. Έως ε, καταναλώτρια με ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα των νανοηλικών, τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν περαιτέρω, α, περισσότερο τουλάχιστον από το να επιτρέψουμε την κλωνοποίηση ζώων. Αυτά είναι τα προβλήματα λοιπόν που μου προκάλεσε η εν λόγω νομοθεσία. Είναι το ζήτημα των κλωνοποιημένων ζώων όχι για επιστημονικούς λόγους αλλά για δεοντολογικούς δεν νομίζω λοιπόν πως αυτό θα πρέπει να είναι και το οριστικό μας επιχείρημα για να εγκρίνουμε ή όχι αυτή την ε, νομοθεσία. Λοιπόν, αντί να τα απαγορεύσουμε, προτείνω να υπάρξει μια ξεχωριστή νομοθεσία και ο Επίτροπος δεσμεύθηκε το να παρουσιάσει μια μελέτη και μια πρόταση. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο πλέον λογικό που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Äh, äh, äh, Κύριος ότι έχει τώρα στήσει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, η δική μας η συγκεντρία δεν ήταν σε θέση να βρίσκεται εδώ, γι' αυτό και θα πάρω εγώ το λόγο. Η δική μας λοιπόν πολιτική ομάδα δεν συμφωνεί με τη θέση του Συμβουλίου, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη ε, τις ανησυχίες που είχε εκφράσει κατά την πρώτη ανάμεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ε, ζώα, καθώς έχει ζητηθεί τόσο αυτά τα ζώα όσο και από γονέντους να μην περιλαμβάνονται, να εξαιρούνται δηλαδή και μάλιστα είχε προταθεί να υπάρξει μια νομοθετική πρόταση να απαγορευτεί η χρήση αυτού του κρέατος. Άρα λοιπόν ε, δεν ε, ε, συμφωνούμε, αλλά η κυρία Σάμπου θέλει να πάμε λίγο ακόμα πιο πέρα από τα όσα είχαμε προτείνει για την πρώτη ανάγνωση, δηλαδή θέλει να, να προτείνει απαγόρευση γενική. Και επίση ε, εκεί σε αυτή την απαγόρευση περιλαμβάνεται η απαγόρευση αυτού του κρέατο από κλωνοποιημένα ζώα και από τρίτε χώρε. Εμεί θα θέλαμε να ακούσουμε τι ε, απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Η δική μα στιώδη υποστηρίζει τη γενική προσέγγιση τη κυρία Ελιοτάρ και την επανεισαγωγή εδώ ε, στο κείμενο των τροπολογιών που είχαμε υποβάλει κατά την πρώτη ανάγνωση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ερικοτοθεσία των γενικά τροποποιημένων, αξιολόγηση κινδύνου νανοτεχνολογιών και ούτω Ευχαριστώ. Ε, ε, Κύριε Στάς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί θεωρώ ότι και στην πρώτη ανάγνωση έκανε ήδη πολύ καλή δουλειά και συνεργάστηκε πραγματικά εξαιρετικά με όλες τις ομάδες και η διάθεση που επικράτησε κατά την πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια αποτέλεσε σαφές αποτέλεσμα της συνεργασίας. Ε, φυσικά δεν μπορούμε να συνταχθούμε απόλυτα με το Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι μας προσέγγισε σε κάποιο βαθμό το Συμβούλιο, αλλά σε ό,τι αφορά τη δική μας ομάδα των Πρασίνων παραμένουν τρία θέματα. Η κλωνοποίηση των ζώων, πολλά χρειάστηκαν να γίνουν στον τομέα αυτό και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την προσέγγιση που επιλέγει η συγγήτρια και όντως είμαστε υπέρ της απαγόρευσης. Θέλουμε ξεχωριστή νομοθεσία. Τα δύο άλλα θέματα για την νανοτεχνολογία υποστηρίζουμε την ε, τροπολογία υπαριθμών 81 της εισηγήτριας. Έκανε ένα βήμα προς το μέρος μας στο Συμβούλιο, θετικό αυτό, και Τρίτο θέμα είναι η επισήμανση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Συμπεριλήφθηκε και σε άλλες νομοθεσίες αυτό, αλλά νομίζω ότι με την τροπολογία υπαριθμών 82 της εισηγήτριας μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε εκ νέου, αν θέλετε, την θέση που είχαμε υποστηρίξει και κατά την πρώτη ανάγνωση. Άρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα των Πρασίνων πρέπει να πω προς την εισηγήτρια ότι θα υποστηρίξουμε την προσέγγιση που προτείνει και δεν θα υποβάλουμε πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Οι υπόλοιποι ομιλητές. Ο Πίτερ Λίζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα της κλανοποίησης ε, των ζώων είναι το πιο σημαντικό το οποίο καλούμαστε να συζητήσουμε, γιατί στα υπόλοιπα θέματα λίγο πολύ η κοινή θέση είναι αποδεκτή να τονίσω κάτι το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα. Φυσικά, υπάρχει εκτροφή ζώων, καλλιέργεια φυτών, αλλά νομίζω ότι όταν μιλάμε για προστασία των ζώων, είναι ευρέως αποδεκτό ότι μιλάμε για κάτι διαφορετικό από όταν μιλάμε για την προστασία των φυτών. Όταν μιλάμε για προστασία των φυτών, μιλάμε για την προστασία ενός φυτού από φυτοφάρμακα, ενώ στα ζώα μιλάμε και για την ε, αποτροπή, αν θέλετε, της ε, κακής μεταχείρισης του ζώου, να μην υποφέρει το ζώο. Αυτό είναι το θέμα, να μην υποφέρει το ζώο. Αυτό αποτελεί ευρωπαϊκό και εκθυμένο στην νομοθεσία και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο πιο πολύ σε βάθο το θέμα της προστασίας των ζώων από ό,τι έκανε το Συμβούλιο. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διοργανώσει μια τέτοια ομάδα διαβούλευσης ε, για την βιοτεχνολογία και η ομάδα αυτή δεν ε, είναι ιδιαίτερα συντηρητική ή κριτική προς τα επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά παρόλα αυτά τοποθετήθηκε κριτικά πολύ εκδικά, επικριτικά σε ό,τι αφορά την κλωνοποίηση αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής ε, Γεωργίας το 2008 με τον, ε, ε, με τον εισηγητή Πάρης και με την έκθεση της κυρίας Λίοταρτ αποφάνθηκε σαφέστατα υπέρ της απαγόρευσης, της γενικής απαγόρευσης, της κλωνοποίησης των ζώων και της εισαγωγής προϊόντων τροφίμων από τα ζώα αυτά. Γενική απαγόρευση, ευρύτατη. Μετά από διπλή συζήτηση, όπως σας είπα. Φυσικά τώρα το θέμα είναι πώς θα το εφαρμόσουμε αυτό στην πράξη. Δεν είναι απλό το θέμα αυτό, ξέρετε. Θα πρέπει να το εξετάσουμε με προσοχή. Ο επίτροπο στην Ακρόαση ανακοίνωσε ήδη ότι πρόκειται να υποβάλει σχετική έκθεση και νομίζω ότι μπορούμε να επιταχύνουμε και την σχετική νομοθεσία, αν δεν υπάρξει μόνο μία έκθεση, αλλά συγκεκριμένη νομοθεσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΜΠΟΕ. Είναι ε, ασαφές. Φυσικά θα ταχθεί υπέρ μίας γενικής ε, απαγόρευσης. Αλλά θα συμπεριληφθεί και ένα απόσπασμα όπου θα αναφέρεται ότι αν θα υπάρξει ζήτημα με την γενική ιδεολογία που επικρατεί στο ευρύ κοινό, θα μπορεί να υπάρξει απαγόρευση. Και αυτό θα το υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα το αποδεχτούν όλα τα μέλη του ΠΟΕ αυτό, αλλά σίγουρα θα άξιζε το κόπο γιατί θα ήταν καλό για όλο την προστασία των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είπε η κυρία Γιούζο ότι υποστηρίζει την προσωπική της άποψη. Εγώ αυτά που λέω τα βασίζω σε δύο ψηφοφορίες που είχαμε στο ΕΛΚ για την έκθεση Πάρης και Λίοταρτ και τουλάχιστον τώρα μετά την ψηφοφορία συζητήσαμε και με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργίας και θα πρέπει φυσικά να δημορφωθεί και η τελική θέση του L, αλλά έχω την εντύπωση ότι κλείνουμε προς την υποστήριξη της θέσης της κυρίας Λίοτάρτ. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει όμως συγκεκριμένες εργασίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλές φορές έχει καλέσει το Κοινοβούλιο την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση. Το έχει υποσχεθεί άλλωστε και η Επιτροπή και θεωρώ ότι το, όλο πρόβλημα της, του κανονισμού για τα τρόφιμα θα επιληθεί σε λίγες μέρες αν ξεκινήσει να δουλεύει το δυνατόν πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποβάλει σχετική πρόταση. Τώρα το ποια θέματα θα συζητηθούν, αυτό θα το αποφασίσει το Κοινοβούλιο με το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά να πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κατά μεγάλη πλειοψηφία, 23 από, τα, 23 από τις 27 χώρες ζήτησαν μια ξεχωριστή πρόταση. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να τηρήσει την υποσχέση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποβάλει και ξεχωριστή πρόταση. Ευχαριστούμε τον Πενταρλίζα. Ο Ρίχαρτ Τζέμπερ τώρα. Για να δούμε τη θέση του ΕΛΚ. Να μην έχουμε μια συνολική άποψη. Ναι, Πρόεδρε, μέσα στο ΕΛΚ είμαστε πολλοί δημοκράτες, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ε, εδώ βέβαια στο συγκεκριμένο σημείο μπορώ να συμφωνήσω πλήρω με τον περιεχόμενο των όσων είπε ο Πέτερ Λίζ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κλωνοποίηση και τα ζητήματα ηθική εκεί, όπω και σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων. Αλλά συμφωνώ και από την οικονομική πτυχή με την θέση του Πέτερ Λίζ για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ε, θα πρέπει να παίξει εδώ ένα διεθνή ρόλο στην παγκόσμια αρένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα είπε ο συνάδελφο ε, Πέτερ Λίζ. Το άλλο τώρα μεγάλο θεματικό πεδίο είναι τα νανοηλικά γιατί εκεί τα ζητήματα, αν θέλετε, τεχνολογικής φύσης είναι ακόμα πιο μεγάλα, ακόμα πιο σημαντικά σε σχέση με την κλωνοποίηση. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να ε, επιτύχουμε περισσότερη πρόοδο ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια ε, του καταναλωτή. Θα πρέπει εδώ να ισχύσει, να εφαρμοστεί η αρχή της πρόληψης γιατί ε, ό,τι κάνουμε εδώ θα πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Ε, και να μην ε, ε, κινούμαστε υπερβολικά γρήγορα σε υλικά τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναλυθεί και αντίστοιχη δράση από την πλευρά της Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί αυτή η ασφάλιση. Μετά ένα τρίτο ζήτημα είναι η έδιγετοθεσία. Η σήμανση είναι λοιπόν ανασφαλίσει οι καταναλωτέ σε ό,τι αφορά την ε, κατανάλωση αυτών των τροφίμων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σαφή ετικετοθεσία για να γνωρίζουν οι καταναλωτέ ότι μπορούν να προβούν στην επιλογή την οποία επιθυμούν και να γνωρίζουν δηλαδή ποια είναι τα τρόφιμα τα οποία α, λαμβάνουν. Οπότε α, αναμένω με ενδιαφέρον ε, αυτά τα όσα έχει υποσχεθεί ότι θα πράξει η νέα επιτροπή γιατί πραγματικά έχουν συγκεντρωθεί μία σειρά, έχουν συσσωρευτεί μία σειρά από νομοθετικέ προτάσει οι οποίε εκκρεμούν. Άρα λοιπόν ε, ε, ελπίζουμε πραγματικά να ενισχύσει λίγο εδώ τι προσπάθειε τη η νέα Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα κείμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μια σειρά ζητημάτων. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ απόλυτα με την θέση της εισηγήτριας που είναι αντίθετη με την ε, χρησιμοποίηση τροφίμων πρόβλημα από κλωνοποιημένα ζώα και από γόνους τους. Αλλά εμπεστός θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα αλλά και στο θέμα των ε, νανοηλικών ε, Είμαι απόλυτα σύμφωνος με την συγκίτρια. Θα πρέπει να αναφέρονται στις ε, σημάνσεις και τα προϊόντα που πρόκειται από τρίτες χώρες επίσης. Θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλους ελέγχους. Θα ήθελα να προσθέσω όμως εδώ και μια κάποια ανησυχία μας. Ε, θα ήθελα η συγκίτρια και η Κομισιό να μου απαντήσουν σχετικά. Και αναφέρομαι στην τροπολογία υπαρθμών 29 που είναι θέση του Συμβουλίου του Συμβουλίου αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα που από τρίτες χώρες εάν αυτά αναφέρονται στον ε, κατάλογο των ε, προϊόντων που από τρίτες χώρες, τότε η εισαγωγή τους θα πρέπει να επιτρέπεται με, ε, σύμφωνα με τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις που γίνεται για τα ασφαλή τρόφιμα. Εδώ όμω με εκπλήσει που δεν αναφέρει, γίνεται αναφορά στα προστατευμένα είδη. Σκέφτομαι την ε, παραδοσιακή χρήση ε, του κρέατος χελωνών ε, που βλέπω που πάει στο Χονγκ βλέπει να χελώνε χελώνες για διατροφή. Υπάρχουν υπάρχουν τα, κάτι άλλο, τα, τα χελιδόνια, τα θέμα της ε, χρήσης ε, κάποιων ε, δοντιών ή άλλων στοιχείων της, ή άλλων τμήματων των τίγρεων. Εκεί είναι, υπάρχει παράδοση χιλιετίας, αλλά στις χώρες μας αυτά τα πράγματα απαγορεύονται. Λοιπόν, μια θέση του Συμβουλίου θα πρέπει να διευκρινίσει το ζήτημα αυτό, διότι θεωρώ απαράδεκτο να μπορούν να ξεπερνούν συγκεκριμένους ελέγχους ή ήδη τα οποία θα απαγορεύονται στην ε, χώρα, στις χώρες μας, διότι υπάρχουν υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στις τρίτες χώρες και οδηγούν στην εξαφάνιση ε, διάφορων, διάφορων ζώων και όχι μόνο, αλλά και φυτών. Ε, και κάτι ακόμα, τροπολογία 25. Και εδώ θα ήθελα την άποψη της Κομισιόν και μια διευκρίνηση την τροπολογία του πολλές φορές μπορεί η μεταφράση να οδηγούν σε παρανόηση. Μιλάμε για πειράματα σε ζώα. Συμφωνώ απόλυτα ότι τα πειράματα επί των ε, σπονδυλωτών θα πρέπει να ε, γίνεται μόνο σε επιπτώσει έκτακτης ανάγκης ε, αλλά όποιος γνωρίζει λίγο από ιατρική γνωρίζει πως, πως ορισμένα πειράματα θα πρέπει να γίνουν επί ζώων που προσωμιάζουν με τον άνθρωπο διότι θα χρησιμοποιούσαμε φάρμακα που θα είχαν και θανατηφόρο ενδεχόμενο αποτέλεσμα στους ανθρώπους, κάτι το οποίο δεν ε, επιθυμούμε. Αυτό που με απασχολεί και με ανησυχεί είναι, ότι ο κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα επιράματα επί σπονδυλωτών θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και να αποφεύγονται οι, ζυπλές, οι ε, ε, πειραματισμοί και πειράματα. Αυτό τι σημαίνει ότι ανεξάρτητα εργαστήρια να κάνουν το ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή να προκαλούν πόνο σε ζώα διότι πρόκειται για πειράματα τα οποία επαναλαμβάνονται. Ναι, συμφωνούμε ότι αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται ή δεν πρέπει να υπάρξει διπλός, διπλό πείραμα κάτι στο ίδιο, επί του ιδίου ζώου, κάτι το οποίο ζητάνε πολλές οργανώσεις προστασίας των ζώων, διότι μερικές φορές είναι απαραίτητο να επαναληφθεί στο αυτό ζώο τα ίδια πειράματα, διότι και έχω υπόψη μου τα νέα συστήματα χημειοθεραπείας ε, το πρόβλημα δεν ε, αφορά την πρώτη, τη δεύτερη χορήγηση του φαρμάκου, αλλά αφορά και συνδέεται σε μια σειρά χορήγησης ε, του φαρμάκου στο ίδιο ζώο και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, διότι η σώρευση αυτού του φαρμάκου μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ε, αντιδράσεις και να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Αν λοιπόν εμείς ζητήσουμε να απαγορευτούν αυτού του είδους τα πειράματα, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να γνωρίζουμε σε περίπτωση που αυτό το σύστημα εφαρμοστεί στον άνθρωπο ποια είναι η αντίδραση του ανθρώπου στην δεύτερη, τρίτη, τέταρτη χορήγηση του φαρμάκου σε περίπτωση υποτροπής. Γι' αυτό λοιπόν ας ε, προσέξουμε πολύ για να απαγορεύσουμε κάτι τέτοιο, διότι δεν θα ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε περίπτωση υποτροπής επαναλαμβάνω ενός ε, καρκίνου επί του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να, ε, για να θέσουμε μια τέτοια απαγόρευση. Αυτά είναι τα δύο ζητήματα λοιπόν, τα πιο σημαντικά, αυτό που συνδέεται με εισαγωγές από τρίτες χώρες των παραδοσιακών προϊόντων, τι σημαίνει κάτι τέτοιο, και η ε, απαγόρευση της ε, διπλής χρήσης, της επανάληψης λοιπόν των πειραμάτων στο ίδιο ζώο, το, κάτι το οποίο λοιπόν αν δεν συμβεί μπορεί να έχουμε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Ευχαριστώ. Θα ενημερωθούμε από τον ε, Έρικ Πουλέ τώρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Διευθυντή της Γενικής ε, Διεύθυνσης ε, Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή, ΣΑΝΚΟ. Θα μας πει λοιπόν σχετικά με το ιστορικό του κλωνοποιημένου κρέατο ε, και τι νομοθετικέ πρωτοβουλίε, ε, τι διπλέ διπλές δοκιμές, double testing, ε, τα ανανοηλικά. Ακούσατε τα όσα θύχθηκαν. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να απαντήσω στις διάφορες πανεμβάσεις που έθιξαν την θέση του Επιτρόπου Νταγή. Θα θυμίσω ότι η διάρκεια της ακρόασης είχε υποσχεθεί πως ε, μια έκθεση θα προτεθεί από την Ευρωπαϊκή Τροπή στο Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο στα τέλη του 2010 σχετικά με την κλωνοποίηση. Επιθυμεί να διατηρήσει φυσικά και αυτήν την υπόσχεσή του και βρισκόμαστε σε φάση διαβούλευσης και τα μέλη της Επιτροπής σας ε, φυσικά θα συναντηθούν με τον Επίτροπο προκειμένου να ακούσει την γνώμη τους. Τώρα βρισκόμαστε λοιπόν, είπα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης των ενδιαφερομένων μερών. Φυσικά η Επιτροπή σας ή κάποια από τα μέλη υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στον τομέα της τροφικής αλυσίδας, επιστήμονες και άλλοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε γύρω στα τέλη του ε, της Ανοίξεως ε, ε, μέσα Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή. Λοιπόν, η έκθεση αυτή θα περιέχει και μια νομοθετική πρόταση, αυτό ακόμα δεν έχει οφασιστεί Θα εξαρθεί από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που έχουν ξεκινήσει ήδη και θα ολοκληρωθούν στα τέλη Ιουνίου. Ε, φυσικά η έκθεση αυτή θα αναφέρει την κατάσταση που κρατεί στον τομέα των κλωνοποιημένων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός ε, των ζώων. Ε, πρόκειται για βοηθοί είτε για ύπους. Είναι ζώα τα οποία έχουν μεγάλη γενετική σημασία, είναι ζώα που χρησιμοποιούνται στους αγώνες, δεν προέρχεται ζώα τα οποία προ... Ε, πρόκειται να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα. Αλλά γνωρίζετε και την άποψη της Κομισιόν ότι δηλαδή μόνο τα κλωνοποιημένα ζώα θα πρέπει να θεωρηθούν ως νέα τρόφιμα και η Κομισιόν δεν συμφωνεί με την άποψη του Συμβουλίου ότι δηλαδή να θεωρήσουμε ως νέα τρόφιμα όχι μόνο τα κλωνοποιημένα τρόφιμα αλλά και αυτά που προέρχονται από την πρώτη γενιά δηλαδή τα τέκνα αν θέλετε τους απογόνους των κλωνοποιημένων κομισιών δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη διότι αυτή η πρώτη γενιά προκύπτει από μια μέθοδο αναπαραγωγής που μπορούσαμε να ονομάσουμε συμβατική είτε με τεχνητή γονιμοποίηση είτε με φυσική γονιμοποίηση. Εμείς η θέση μας ήταν σαφής, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κλωνοποιημένα ζώα ως ε, νέα ζώα τα οποία θα πρέπει να περάσουν από την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων. Τώρα για τα νανο, νανοτεχνολογίες ε, τώρα στο σχέδιο κανονισμού που συζητάτε Φυσικά υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος προέκυψε από την πρώτη ανάγνωση, διότι δεν υφίστατο στην αρχική πρόταση της Κομισιόν του Ιανουάριου 2008. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι τεχνολογίες εξελίσσονται τάχιστα και σε επίπεδο Κομισιόν με ορισμένες ε, ε, εμπλεκόμενες γενικές διευθύνσεις περιβάλλοντος, έρευνας, ε, βιομηχανίας, ε, επιχειρήσεων κλπ. Να ζητάμε από την Επιστημονική Επιτροπή να οριστικοποιήσει έναν ορισμό των νανοτεχνολογιών που θα πρέπει να είναι απλός και εφαρμόσιμος, δηλαδή να μπορεί να ελέγχεται από τις αρχές των κρατών μελών τόσο όταν υπάρχουν ε, προϊόντα νέων τεχνολογίες που ε, μπαίνουν στην ε, τροφική αλυσίδα, όσο και υλικά τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας νομικός ορισμός αλλά και να υπάρξουν και τα κατάλληλα μέτρα σε επίπεδο εργαστηρίων για να ελέγχουν αυτόν τον ορισμό τότε είναι ένας ορισμός ο οποίος δεν έχει συνέπεια αναφορικά με τον έλεγχο και τους ελέγχους που πρέπει να ασκούνται. Επιθυμούμε λοιπόν να είναι εύκολα επαληθεύσιμο από τις ελεγκτικές αρχές έτσι ώστε να απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία πρόκειται από τεχνολογίες αλλά δεν έχουν δηλωθεί ως διούτα και Εδώ προκύπτει και το ζήτημα της επισήμανσης και πληροφόρησης των των ε, καταναλωτών. Ξέρετε ότι επίπεδο καλλιντικών ε, υπάρχει μια ρύθμιση για το ζήτημα της επισήμανσης. Όταν χρησιμοποιούμε ένα καλλιντικό το οποίο περιέχει νοοτεχνολογίε, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στα περιεχόμενο, στα συστατικά του προϊόντος και αυτό αφορά και στα τρόφιμα, αλλά με την προϋπόθεση, επαναλαμβάνω, να είναι κάτι το οποίο θα είναι ελέγξιμο και επαληθεύσιμο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του κράτους μέλους. Για να απαντήσω στην παρέμβαση του κυρίου Ρώση για το ζήτημα του κρέατος της χελώνας από το Χονγκ Είναι προφανές ότι τα τρίτες χώρες θέλουν να εξαγάγουν τρόφιμα τα οποία προέρχονται από ζώα που προστατεύονται με βάση τις ήτες, δηλαδή την σύμβαση που προστατεύει τα υποξαφάνιση ζώα και φυτά. Αυτά τα προϊόντα λοιπόν που προέρχονται από τα, τα ζώα δεν μπορούν να εισαχθούν. Αποκλείεται λοιπόν να ε, φάμε ε, ένα κρέας από, κρέας από χελώνα, εφόσον αναφέρεται στην ε, κατάλογο της σύμβασης του ε, ΣΥΤΕΣ, ε, μπορεί λοιπόν, εφόσον θα έχει ελεγχθεί από την ΕΦΣΑ και να θεωρηθεί ως νέο προϊόν, νέο τρόφιμο. Εάν είναι προστατευόμενο λοιπόν το είδος, το κρέας, τα αυγά κλπ ή και οι τρίχες δόντια από την ε, τίγρεως ε, δεν μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν σε τρόφιμα. Τώρα, σε ό,τι φορά τα πειράματα επιζών, γνωρίζετε πως η Κομισιόν έχει συντάξει νομοθεσία βασισμένη στον κανόνα των τριών R στα αγγλικά, replaced, restricted και refined. Δηλαδή, κάθε πείραμα σε ζώο θα πρέπει να αντικατασταθεί σιγά σιγά από εναλλακτικές μεθόδους που δεν ε, θα ε, χρησιμοποιούν την ε, ζώα είτε πρόκειται για ποντίκια, μην μιλήσουμε για πυθίκους και σκυλιά. Θα υπάρχουν λοιπόν αυτές οι εναλλακτικές μέθοδοι οι οποίες δίνουν ισοδύναμα αποτελέσματα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ζώντα, ζώα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα το οποίο η Κομισιόν ε, έχει δεσμευθεί και υπάρχουν πολλές ε, κανονιστικές διαδικασίες ε, για να καταργήσουμε αυτά τα πειράματα σε ζώα και μία από τα τελευταία αφορά τον έλεγχο των ε, οστράκων ε, όπου χρησιμοποιήσαμε ε, ποντίκια για να δούμε κατά πόσον δεν περιέχουν τοξίνες κλπ. Τώρα αυτά τα πειράματα αντικαθίστανται από χημικές μεθόδους. Φυσικά υποστηρίζουμε τις τροπολογίες που επιθυμούν να περιοριστούν η χρήση ζώων σε πειράματα, διότι αυτό επισέρχεται σε ένα πρόγραμμα που ισχύει εδώ και κάποια χρόνια αναφορικά με τον περιορισμό της χρήσης ζώων στα πειράματα. Αυτά, Πρόεδρε, μπορεί να σας πει η Κομισιόν σε αυτή την φάση. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπουλέγκα τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Νομίζω πως η φιλελεύθερη δεν πήραν τον λόγο. Ίσως ε, ο Θαλής νομίζω από το Παρίσι σήμερα έχει μια καθυστέρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην συνάδελφο πρωτού επιτρέψουμε στην συγγήτρια να ξαναμιλήσει. Α, όχι και ο Έρχαρντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά ε, υποστηρίζω την εξαιρετική έκθεση της κυρίας Ντοτάρ με την οποία επανειλημμένα συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα εδώ οι τι τεχνολογίε. Όντως είναι παρούσε σε πολλά προϊόντα, αλλά δεν γνωρίζουν ποια είναι τα σχετικά προϊόντα, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη έγκριση και ούτε επισήμανση τώρα εξολόγηση του κινδύνου είναι ανεπαρκή, νομίζω ότι το τονίστηκε και πως πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν τους κινδύνου που υπάρχουν ε, κάποιε που προκύπτουν από τη χρήση κάποιων ε, νανοτεχνολογιών και νανοηλικών. Νομίζω ότι θα πρέπει να βασιστούμε στην ε, προηγούμενη εμπειρία μας και να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ανησυχία μας για το, το Συμβούλιο δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του και διότι α, θέλουμε να χρησιμοποιήσουν τέτοιες τεχνολογία θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες ε, έρευνες και εγκρίσεις. Τώρα η κλωνοποίηση, η κλωνοποίηση δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και δημιουργεί πόνο στα ζώα. Το Συμβούλιο θέλει να αποκλείσει την ε, να ρυθμίσει το των εκλογμένων ζώων και του απογόνου ε, για να μην υπάρχει ένα νομικό, ε, ε, νομικό κενό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει τάχιστα μια πρόταση η οποία θα καλύπτει όλε τι πτυχέ τη κλωνοποίηση. Και θα κλείσω, Πρόεδρε με κάτι το οποίο συνεχώ επαναλαμβάνω που είναι η προστασία του πλουραλισμού, δηλαδή η εφαρμογή του, της αρχής της προστασίας ε, είναι κάτι το απαραίτητο. Ε, διαφάνεια θα πρέπει να έχουμε δεδομένα τα οποία να δημοσιεύονται και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια όπως επανειλημμένα ζήτησε το Ευρωπαϊκή ο ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο χρειαζόνται γνωμοδοτήσει των εμπειρογνωμόνων από όλες τις πλευρές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τρόπο ευφυή για την εμπειρογνωμοσύνη. Θα πρέπει να υπάρχει και εδώ μια συνεργασία με τα κράτη-μέλη, να λαμβάνει η ΕΦΣΑ υπόψη της, ε, της θέσης τους. Ε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα περιβαλλοντικά και να μην αφήνει τα θέματα αυτά μόνο στην ΕΦΣΑ και να μην ξεχνάμε πρόεδρα πως αυτές τις ε, περιόδους ε, που διανύουμε το ζήτημα της ηθικής και της διοντολογίας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποια πολύ σύντομα ε, σχόλια να κάνω. Καταρχήν να πούμε ότι υποστηρίζουμε τη θέση του Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε εδώ να, να αναμένουμε μια πολύ σαφή νομοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση με αυτή την πρόταση τα δικαιώματα που σχετίζονται με την προστασία των ζώων πράγματι θα έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να τα επιβάλλουμε έναντι του Συμβουλίου. Εάν όμως για αυτά τα προϊόντα επιθυμούμε μια επιπρόσθετη εδώ νομοθεσία, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και για άλλα προϊόντα ε, διαφορετικές νομοθετικές πράξεις όπως για γενετικά τροποποιημένα υλικά. Δηλαδή η τροπολογία 18 η οποία ε, ζητάει να υπάρχει ετικετοθεσία ε, για ζώα τα οποία έχουν τραφεί με ζωοτροφές από γενετικά τροπημένους οργανισμούς ε, δεν έχει θέση εδώ καθώς ήδη αυτό καλύπτεται από άλλη σχετική νομοθεσία δική μας που ήδη υπάρχει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένας σωστός συντονισμός και μια αποσαφήνιση και μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Σε ό,τι αφορά την ανοτεχνολογία τώρα. Ε, Κυρίε και κύριοι, θεωρώ πω πρόκειται για μια πολύ σημαντική τεχνολογία η οποία μα ε, ανοίγει πολλέ δυνατότητε και θα ήθελα να παρακαλέσω να μην ξεκινήσει μια συζήτηση σε καθεστώ πανικού για μία ακόμα φορά ως προς τους κινδύνους, ως προς τις αντικέ συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν. Προφανώς και θα πρέπει να διαρευνηθούν όλα αυτά. Προφανώς και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά το να γίνονται από τώρα συζητήσεις ως προς το πόσο επικίνδυνα είναι όλα αυτά ε, δεν έχει ε, νόημα. Μιλάμε δηλαδή για προϊόντα στα οποία έχει μεταβληθεί αν θέλετε το μέγεθος ε, των μορίων. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως ε, θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι και λίγο πιο επικοδομητικοί στη συζήτηση που θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά και πάλι το λόγο. Κύριε Πουλέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ολοκλώσω την ε, παρέμβαση κυρία Λεπά σχετικά με τις νανοτεχνολογίες που ανέφερε ότι περιέχονται σε πολλά προϊόντα. Είναι γεγονός ότι οι νανοτεχνολογίες ε, αφορούν τις ε, καινοτομίες, υπάρχει μεγάλη ζωτικότητα στις βιομηχανίες και στα βιομηχανικά προϊόντα χρησιμοποιούνται, όπως π.χ. όλα τα ελαστικά των αυτοκινήτων γίνονται με προϊόντα περιδών τεχνολογίας. Αλλά στα τρόφιμα, σύμφωνα με τις προφορίες που λάβαμε από τις Εθνικές Αρχές των 27 κρατών μελών και από τις ε, βιομηχανίες ε, κατασκευής τροφίμων, ε, δεν υπάρχουν ε, τέτοιες ε, τεχνολογίες στην, ε, στην κοινωνική αγορά. Υπάρχουν στις Ηνωμένε Πολιτείε ιδιαίτερα, αλλά για μας είναι σαφές πως τα προϊόντα αυτά, ακόμα και αν δεν υπάρχει ορισμό στον προηγούμενο κανονισμό για τα νέα τρόφιμα, οι τεχνολογίες όταν εισάγονται στα τρόφιμα τροποποιούν ουσιαστικά τα συστατικά τους ε, και δεν υπήρχαν πριν το 97 και τα εμείς θεωρούσαμε ότι πρόκειται για νέα τρόφιμα και θα χρειαστεί να αξιολογηθούν από την ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων και μπορούμε ως εκ τούτου να δηλώσουμε ότι στην κοινωτική αγορά δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ε, τρόφιμα υπάρχουν τρόφιμα που, ε, που κατασχέθηκαν στα σύνορα ε, προελεύσεως ε, από τρίτες χώρες αυτά τα τρόφιμα επαναπροωθήθηκαν στην χώρα προέλευσης και έχουμε μια λογική βεβαιότητα διότι δεν μπορεί η Κομισιόν να τα ελέγχει όλα και να τα γνωρίζει τα πάντα αλλά Είμαστε βέβαιοι ότι στην κοινότητα, στις αγορές της κοινότητας δεν υπάρχουν τέτοια τρόφιμα. Είναι μια διευκρίνηση που θα ήθελα να κάνω. Ναι, όντω όταν ε, η Επιτροπή μετέβησε στην Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο, ακούσαμε ότι η νοτοκτολογία στη ΣΥΠΑ θεωρείται ως η τεχνολογία του μέλλοντος και προωθείται σε όλα τα επίπεδα θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν στην Ευρώπη τι ακριβώς κάνουμε, κατά πόσον ε, ενέχονται κίνδυνοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΕΦΣΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις σχετικές επιστημονικές ε, ενδείξεις. Κυρία τα ακούσατε τα σχόλια και τώρα παρακαλώ η τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες εισηγητές αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής να τους ευχαριστήσω ασφαλώς και για την καλή συνεργασία κατά την πρώτη ανάγνωση. Είδαμε ότι επικρατεί γενικά μια συνένεση στο Κοινοβούλιο. Δεν ακούω αντιφατικές ιδιαίτερα απόψεις. Όλοι λίγο πολύ υποστηρίζουμε αυτά που αποφασίσαμε το 2008. Με ικανοποιεί λοιπόν αυτή η διαπίστωση και θεωρώ ότι πρόκειται για μια σωστή βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω μ, τη βοήθεια όλων των σκιωδών αλλά και των υπόλοιπων μελών, γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητο το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή, γιατί, όπως είπαμε, είναι ταχαίως αναπτυσσόμενος ο κλάδος της νανοτεχνολογίας. Θα θέλαμε να υπάρξει μια λύση και για την ε, κλωνοποίηση και για τα νέα μέσα στην τεχνολογία των τροφίμων. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική. όταν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχουν ακόμα στην αγορά προϊόντα με νανοτεχνολογία. Κοιτάξτε, δεν θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση αυτή, αν με διαβεβαιώνετε ότι έτσι είναι τα πράγματα, εντάξει το δέχομαι, αν και έχω κάποιες αμφιβολίες. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να παραμείνει η κατάσταση έτσι έως ότου έχουν γίνει οι απαραίτητοι Έλεγχη ασφάλειας για τον καταναλωτή. Και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Να υποδείξω ωστόσο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο ρόλος που παίζει είναι ρόλος κλειδί. Γιατί, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί με συντριπτική πλειοψηφία ότι θέλει διαφορετική νομοθεσία για την κλωνοποίηση των ζώων και για την διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυτών. Αν διτηθούν καν στην αγορά τα προϊόντα αυτά των κλωνοποιημένων ζώων και αυτό θα πρέπει να τεθεί και στο ευρύ και πολλά κράτη-μέλη έχουν υποδείξει και αυτά ότι θέλουν ξεχωριστή νομοθεσία για την κλωνοποίηση και ότι ελπίζουν να μην προκύψει χάσμα στην νομοθεσία και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η τοποθέτηση ως σημείο εκκίνησης δεν είναι σωστή. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει κατεπηγόντως μία πρόταση σε ό,τι αφορά την κλωνοποίηση των ζώων προκειμένου να κάνουμε και μεγάλα βήματα προόδου σε ό,τι αφορά άλλε νομοθεσίε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ενοτεχνολογία. Θέλω επίση μεγαλύτερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά τι δοκιμέ ε, στα ζώα και ελπίζω να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή τον Ιούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια γνωρίζει το θέμα αυτό ασφαλώς η Επιτροπή μας και είδαμε ότι επικρατεί αρκετά μεγάλη συμφωνία. Θα θέλουμε να προωθήσουμε την νομοθεσία αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντική η νομοθεσία αυτή και για την ε, οικονομική διάσταση. Προθεσμία για τις τροπολογίες 13 Απριλίου, 13 Απριλίου για να ψηφίσουμε το Μάιο στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια. Τα πήγαμε πολύ καλά, λέει ο Πρόεδρος, γιατί ο επίτροπο καταφτάνει στι 11. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να παρακαλέσω τους συναδέλφου να ξαναέλθουν στι 11, γιατί μιλάμε για το πρόγραμμα για το περιβάλλον για την τρέχουσα θητεία. Τα ξαναλέμε λοιπόν στι 11. AUTHORWAVE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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zurück. Αγαπητοί κυρίε και κύριοι, συνάδελφοι, επιστρέφουμε λοιπόν στι εργασίε τη Επιτροπή μα. Στο σημείο 13 τη ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Περιβάλλοντο Γιάννη Ποτότσνικ, τον οποίο καλωσορίζω θερμά σήμερα εδώ στην Επιτροπή μα. Έχουμε ε, πολύ καλέ αναμνήσεις και από την ακρόασή του πριν από την εκλογή δηλαδή της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο. Και καλωσορίζω και τον Καρλ Φάγκεμπεργκ, τον Γενικό Διευθυντή, τον οποίο γνωρίζουμε καλά από όλη την ε, συζήτηση για τις κλιματικές μεταβολές κατά την περίοδο πριν από την Κοπεχάγη. Κύριε Επίτροπε Ποτότσινγκ, σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είχαμε ήδη συζητήσει κάποια ζητήματα στο ε, πλαίσιο της ακρόασης. Έχουν παρένθει τώρα κάποιοι μήνες και γι' αυτό θα θέλαμε βέβαια προφανώς να ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα έχετε προβλέψει για την επόμενη περίοδο στο πλαίσιο των εργασιών σα. Οπότε θα ήθελα να αξιοποιήσουμε την επόμενη μία μισή ώρα που έχουμε στη διάθεσή μα για να συζητήσουμε τα βασικά ζητήματα τη ε, πολιτική ε, για το περιβάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα δίνω λοιπόν ε, το λόγο για την παρουσίασή σα, κύριε Επιτροπή. Thank you, President. Uh, good day to everybody. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εμφανιστώ σήμερα ενώπιον σας όπως ανέφερε ήδη ο Τζο ε, έξι εβδομάδες έχουν περάσει από το ακρόασή μου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Είναι ακόμα νωρίς αλλά ήδη έχει γίνει κάποια πρόοδος σε σημαντικά ζητήματα τα οποία θα σας αναφέρω εντάχει όπως το Ρίτσου και το ζήτημα των ε, ε, ειδών που βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να σας μιλήσω για το όραμά μου για το, σχετικά με το περιβάλλον και το πώς ε, φαντάζομαι να το εφαρμόσω. Επενδύσαμε μεγάλη ενέργεια σχετικά με την πρόθεση της Στατικής Λισαβόνας και χαίρομαι που ε, το Ευρώπη το 2020 έχει συμπεριλάβει την υπερβαρική πολιτική στην, ε, στο πρόγραμμά της. Αυτό νομίζω είναι σύμφωνα με τα όσα επιθυμούν οι Ευρωπαίοι παράλληλα με την αύξηση της ε, απασχόλησης και την οικονομική μεγέθυνση. Μιλήσαμε πολύ στο παρελθόν για την αηφορία και την βιωσιμότητα θα ήταν ε, ανεύθυνο σε καιρούς όπου έχουμε πολύ υψηλή ανεργία και σημαντικά προβλήματα οικονομικής φύσης ε, να μην επικεντρώσουμε προσοχή μας σε ό,τι αφορά την οικονομική μεγέθυνση και την, ε, και την απασχόληση. Αλλά επίσης θα πρέπει να ρωτούμε τι είδους ανάπτυξη επιθυμούμε και τι είδους απασχόληση. Θεωρώ λοιπόν πως το EU 2020 θέτει τα δύο αυτά ζητήματα στο σωστό πλαίσιο. Ε, ο πληθυσμός του πλανήτη το 2050 θα φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα των πόρων. Και αυτό, όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχουμε καμία επιλογή, αλλά από το να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο παραγωγής αν θέλουμε να διτηρήσουμε τον πλανήτη μας σε καλή φόρμα για τις επόμενες γενιές. Χρειάζεται να προωθήσουμε πολιτικές οι οποίες ε, θα έχουν τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι μας για τα προσεχή έτη. Θα ενθυμίσετε στην ακρόασή μου, ανέφερα τις ε, τρεις προτεραιότητές μου να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να ε, κάνουμε πιο δυνατή την οικονομία μας και να ε, διασφαλίσουμε την σωστή χρησιμοποίηση της ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ανέφερα τα προγράμματά μας για θέματα βιοποικιλότητας, τεχνολογιών κλπ. και την αποτελεσματικότητα των, της χρήσης των πόρων. Πρώτα απ' όλα τα προγράμματά μας για το 2010. Η πράσινη ανάπτυξη, όπως ξέρετε, είναι ένα κεντρικό ζήτημα για την πολιτική της Ευρώπης το 2020, αλλά δεν πρόκειται να επιτευχθεί εάν δεν λάβουμε τα σωστά μέτρα. Βιοπικιλότητα αποτελεί μια πηγή πολύ σημαντική για μας, μας παρέχει τα ύδατα, την ξυλία και άλλους πόρους ιδιαίτερα σημαντικούς. Εάν δεν διαχειρίσουμε τα οικοσυστήματά μας θα χάσουμε τμήμα αυτών των πόρων και θα μας κοστίσει ιδιαίτερα ακριβά για να αντικαταστήσουμε αυτούς τους πόρους με τεχνητούς. Παρά λοιπόν τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει μέχρι τώρα, η βιοπικιλότητα μειώνεται διότι παράλληλα υπάρχει και επιτάχυση στην αύξηση του πληθυσμού. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν και η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το ε, όραμα του στόχου και του στόχου στο 2020 είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αποτελεί έναν, ένα κεντρικό τον ε, ακρογωνία λίθο για το μέλλον μας και το πλαίσιο διαπραγματεύσεων που θα γίνουν στην Κοία αργότερα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει με μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Προσβλέπω το να ακούσω τις θέσεις σας ε, πάνω στο ζήτημα αυτό ε, μέσω της έκθεσης ε, κύριε Ντελόγκ. Θα καταβάλω ιδιαίτερες προσπάθειες για να προωθήσω την στρατηγική για τη δύο μετά από τι διαπραγματεύσεις στην Γκόια. Αυτή η στρατηγική αποτελεί ένα τμήμα του προγράμματο ε, για φέτο. <clears throat> Η στρατηγική για την ποικιλότητα θα εξαρτηθεί επίση από τι ε, πρωτοβουλίε που θα αναλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα επικεντρωθούν και θα ε, συμπεριληφθούν σε βασικέ πολιτικέ. <clears throat> Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει από κοινού να συνεργαστούμε τους προσεχείς μήνες. Πάντως ε, προστασία του φυσικού μας, των φυσικών πόρων δεν επαρκούν. Θα πρέπει να προωθήσουμε την πράσινη ανάπτυξη. Αυτό θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα και σε συνεργασία με το θέμα της βιοποικιλότητας. Η οικοβιομηχανία. Είναι ένας ε, από τους πλέον δυναμικούς ε, βιομηχανικούς τομείς ε, στην Ευρώπη. Δημιουργεί θέσεις απασχόλησης σε πολλούς κλάδους, αλλά θα πρέπει να την προωθήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να συμπεριλάβουμε τους τομείς των νέων υπηρεσιών και τις υπηρεσίες στα νοικοκυριά. Πρέπει να προωθήσουμε τις νέες πράσινες τεχνολογίες θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εδώ το παράδειγμα των αποβλήτων που τώρα έχει αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ε, διάθεσης, χρήσης, ανακύκλωσης κλπ. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν καθαρές βιομηχανίες και όχι μόνο να φροντίσουμε να καθαρίσουμε τις ήδη, καθαρίσουμε πιο καθαρές μάλλον τις ήδη υπάρχουσες. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν τις νέες πράσινε τεχνολογίες και στον τομέα των υπηρεσιών. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε αγορές για ζητήματα οικολογικής καινοτομίας, να ανοίξουμε τις αγορές και προς αυτό συμφώνησα με τον Δ. Μάιε Κράμερ που ήταν ε, υπουργό ε, ανάπτυξη στην Γερμανία, τελευταίες δύο κυβερνήσεις και θα είναι και προσωπικός μου σύμβουλος για ζητήματα που άπτονται με το θέμα της ε, οικολογικής καινοτομίας και για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Το 2011 θα εξετάσουμε και περαιτέρω το θέμα της οικολογικής ανανέωσης και καινοτομίας. Θα πρέπει να έχουμε προγράμματα για να καταστήσουμε την Ευρώπη πλέον αποτελεσματική. Αυτά προκύπτει και από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Είναι μία από τι 7 βασικέ πρωτοβουλίε που προτείνουν για την Ευρώπη του 2020. Όλο αυτό συνδέεται με το θέμα της ε, ανάπτυξης, ε, της μεγέθυνσης και της παραγωγικότητας. Δυστυχώς δεν μπορείτε να δείτε αυτό το διάγραμμα. Έχουμε την παραγωγικότητα αφενό και την ανάπτυξη και την απασχόληση ε, στον άλλο στον, στον κάθετο άξονα. και, και κάτι ακόμα. Ε, πρέπει να υπάρξει μια νέα λογική των επιχειρηματιών για το πώς χρησιμοποιούνται οι πρώτες ύλες, οι νέες τεχνολογίες κλπ. Αυτό θα μας καταστήσει πιο αποτελεσματικούς και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να καταστούμε πιο αποτελεσματικοί και πιο αποδοτικοί. Χρειάζεται να προσέχουμε την χρήση των ε, νέων πόρων, των πόρων η μελλοντική γεωστατική μας θέση έχει μεγάλη σημασία και χρειάζεται να ε, σφίξουμε τις ζώνες και να εξορροπήσουμε τα δημοσιονομικά μας. Πρέπει να φροντίσουμε να παράγουμε περισσότερα, αλλά με τρόπο πλέον βιώσιμο. Υπάρχει, προχωράμε στην περίοδο της ε, ανακύκλωσης ε, όλοι οι πόροι, ύδατα, ορυκτά, ε, ξυλία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πιο αποτελεσματικό τρόπο για να πάψουμε να επηρεάζουμε τόσο σημαντικό το περιβάλλον. Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Οι οικονομικές προϋποθέσεις είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Εάν Ε, θα ενθυμίσετε πολύ καλά την ενεργειακή κρίση. Τότε η τιμή των ενέργειας του πετρελαίου ήταν ιδιαίτερα υψηλή και αυτό ε, οδήγησε σε χρηματοδότηση της ε, έρευνας και της ανάπτυξης. Αργότερα οι τιμές μειώθηκαν αισθητά και ζήσαμε μερικές δεκαετίες ψευδέστησης. Αυτές οι δεκαετίες όμως παρήλθαν και αυτό το οποίο μας έχει μείνει είναι τα προβλήματα που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε όπως οι κλιματικές αλλαγές και όλα τα ζητήματα που άπτονται του θέματος αυτού. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι τα μηνύματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πάντα ξεκινάμε από τα βασικά, από τις προφορίες που μας παρέχει το σύστημα. Έχουμε διάφορα εργαλεία για την πνευματική ε, προστασία αλλά υπάρχουν και ζητήματα εγκάρσια, αφορούν πάρα πολλές ε, του ανθρώπου και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις οικονομικές και βιομηχανικές πολιτικές ε, της Ευρώπης. Γι' αυτό και η στρατηγική του 2020 είναι το σωστό εργαλείο για να το πετύχουμε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συνεργαστώ στενά με τους συναδέλφους μου, ειδικά τους επιτρόπους επίθεων για την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία, το εμπόριο, την έρευνα και με τους ε, υπολείπους σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να θέσουμε τις κατάλληλες κατευθύνες γραμμές και να ε, υπάρχουν ε, σωστοί μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου. Φυσικά δεν ξεκινάμε από το μηδέν, έχουμε πολύ καλές πρωτοβουλίες, έχουμε την πρόγραμμα i4 ανάπτυξης, ε, πρωτοβουλίες για τις πρώτες ύλες, Πολλά κράτη-μέλη επίση έχουν να μας δώσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ε, να πετύχουμε συμφωνία για ένα πρόγραμμα ομπρέλα που θα καλύπτει δηλαδή τους παρακάτω στόχους. Μεγαλύτερη αηφορία σε ό,τι φορά την ε, κατανάλωση. Να, ε, αξιολοποιήσουμε τις, τους πόρους μας, ε, να προωθήσουμε το ζήτημα των προμηθειών του δημοσίου με πράσινες ε, τεχνολογίες, να ε, αντικαταστήσουμε τα προϊόντα τα οποία ρηπαίνουν πόρος που είναι απεριόριστος, ευτυχώς, είναι η εγκέφαλή μας και ελπίζουμε να το χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα το 2011. Επίσης βλέπουμε ότι θα είναι και η τελική αξιολόγηση των έξι προ... Ε, πυραβολτικών προγραμμάτων. Θα τα λάβουμε όλα αυτά ως βάση για τις εργασίες που θα προχωρήσουμε το 2012 αλλά και την πρόθεση του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου. 2012 τα προγράμματά μας έχουν αρχίσει να παίρνουν σάρκα και ωστά ήδη από τώρα. Ε, θα επικεντρώσουμε προσοχή μας στο νερό επαρκές και καθαρό νερό είναι απαραίτητο για όλες τις δραστηριότητες. Το 2012 προβλέπω να υποβάλω ένα πρόγραμμα για τα ύδατα της Ευρώπης που θα <clears throat> ζητάει την, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ύδατα και θα εξετάζει επίση και άλλου τομεί που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νομοθεσίε ε, οι οποίε ε, εγκρίναμε τα τελευταία χρόνια για τα αέρα, για τα απόβλητα και για τα χημικά εφαρμόζονται με σωστό τρόπο και να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 υποστηρίζει την πράσινη ανάπτυξη όπως και το επιθυμούσαμε. Ξέρουμε ότι πολλά έχουμε να κάνουμε στον τομέα αυτό ακόμα. Και εδώ θα επικεντρωθώ κυρίως ε, στο να οικοδομηθούν ε, γέφυρες που θα διασφαλίσουν ότι τα κράτη-μέλη είναι δεσμευμένα στα θέματα εφαρμογής προκειμένου να διασφαλίσουμε και την ε, εφαρμογή των μέτρων αυτών, αλλά δεν θα προβώ και σε περιττές τέτοιες ενεργείες. Στην πρώτη μου επίσκεψη στη χώρα μου πριν από 14 ημέρε. πρόκειται για την ακριβή ημερομηνία που ξεκίνησε και η διαδικασία επί παραβάση ε, κατά την ε, χώρα αυτή. Νομίζω ότι ήταν σαφές το μήνυμα λοιπόν. Τα στοιχεία τα οποία επεξήγησα θα συμπληρωθούν και από δραστηριότητε σε άλλου τομεί, όπου χρειάζεται ευρωπαϊκή δράση για να ενισχυθεί η πράσινη οικονομία. Δεν ε, μπορώ να καλύψω όλα αυτά τα θέματα εδώ και τώρα σήμερα, αλλά να σας αναφέρω ορισμένα εξ αυτών. Φέτος θα εξετάσω τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, την νομοθεσία για το πόσιμο νερό σε ό,τι αφορά τα υγρά κάψιμα και τα μεγάλα ατυχήματα, καθώς και αναθεωρήσεις ε, για την χρήση καδμίου σε μπαταρίες και τη σχετική στρατηγική. Στο απότερο μέλλον θα συνεργαστώ για την ε, αναθεώρηση του καταλόγου των προτεραιοτήτων στα πλαίσια της ε, ε, νομοθεσίας για το Natura, για το περιβάλλον και θα χρειαστώ μεγάλη βοήθεια από δική σας πλευράς στο πώς θα πρέπει να αναδιαμορφώσουμε την κοινή αγροτική πολιτική, την κοινή αλληλευτική πολιτική και πώς θα θέσουμε στη σωστή βάση της ε, στη σωστή βάση τους τα συμφέροντά μας κατά την επόμενη δημοσιονομική προπτική. Τέλος, υπάρχουν κάποια νομοθετικά ζητήματα τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη και θα ήθελα να συνεργαστώ και με εσά και με τις Προεδρίες και με το Συμβούλιο. Θα πρέπει το IPCC και η νομοθεσία για την παράνομη να ολοκληρωθούν με επιτυχία για το VEE e επίσης και για τα βιοκτώνα ασφαλώς. Η επιτυχία που θα σημειώσουμε θα εξαρτηθεί όχι μόνο φυσικά από τη δική μου πρόταση, αλλά και από την ε, θέση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Έχουμε τη στρατηγική το 2020 που είναι καλή, αλλά η στρατηγική από μόνη της σίγουρα δεν πρόκειται να αποδώσει καρπούς. Είναι σημαντικό να τράξουμε την ευκαιρία αυτή και να εφαρμόσουμε στην πράξη όλα όσα έχουμε διακηρύξει και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεργαστούμε στενά και πολύ ενεργά. Να μην μείνουμε στα γραπτά, σε αυτά που έχουμε γράψει. Ελπίζω να μπορώ να υπολογίσω στην υποστήριξή σας κατά την προσπάθεια αυτή και το ελπίζω αυτό σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα μέλη της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ. Yeah, Dank, äh, Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε Ποτόσνικ για το όραμα αυτό, τη φιλοσοφία αυτή που μας παρουσιάσατε για την Ευρώπη που θα εξοικονομεί τους πόρους της για το πακέτο αυτό ιδέων και μέτρων τα οποία επίκυνται. Είμαστε πολύ περίεργοι εδώ πέρα στην Επιτροπή. 25 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Να περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στους συναδέλφους Δύο λεπτά να προτείνω γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουν όλοι και οι συντονιστές. Και ο κύριος Ζέμπερ θα ξεκινήσει και θα δώσει το καλό παράδειγμα. Και το νερό ασφαλώς αποτελεί βασικό θέμα. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός ο Επιτροπός και στην ακρόαση και τώρα βελτίωσε ακόμα την ε, παρουσίασή του. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα τις ιδέες σας για το θέμα του νερού Μία συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Επίτροπε. Βλέπουμε τώρα στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για το νερό ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της ε, ε, της υδάτινης ε, αυτής, του υδάτινου δυναμικού. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω μιας γενικής ρύθμισης να δημιουργηθεί ένα ισότιμο επίπεδο για να μην υπάρχουν τέτοιες μεγάλες διαφορές και να μην υπάρχουν τέτοια μεγάλα χάσματα. Ίσως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με εξισορροπητικό ρόλο. Μία άλλη ερώτηση Πολλές καλές ιδέες αναφέρατε, αλλά δεν αναφερθήκατε καθόλου σε θέματα επικοινωνίας. Όπως ξέρετε, η περιβαλλοντική πολιτική χαρακτηρίζεται από πολλά και ωραία οράματα, αλλά χρειάζεται και συγκεκριμένη εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Μόνο έτσι μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες, γιατί πολύ καλές ιδέες σας, αλλά πολλές φορές ο κόσμος δεν θέλει να ακολουθήσει τις ιδέες αυτές. Τι σκοπεύει λοιπόν να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά αυτή την επικοινωνία με το κοινό. Πώς σκοπεύει να διαβιβάσει αυτό το μήνυμα για να μας υποστηρίζει ο κόσμος. Ένα άλλο θέμα είναι γενετικό τροποποιημένοι οργανισμοί. Ξέρω ότι δεν είσαστε εσείς αρμόδιος, αλλά παρόλα αυτά η εκτίμηση του κινδύνου σε ό,τι αφορά τους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς σχετίζεται με το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου και από την πλευρά αυτή να καλυφθείτε. Και για να τηρήσω λοιπόν τα δύο λεπτά θα περιοριστώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Λίντα Μακέβεν. Ευχαριστώ. Επίτροπε, σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα. και έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε ότι θα χρειαστούμε συνοχή τη πολιτική. Ε, μιλήσατε για την ενέργεια. Ε, στην δεκαετία του 70 θέλαμε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργεια. μετά στη συνέχεια ε, πήγαμε στην πιο φθηνή ενέργεια. Και τώρα έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση να χρειαζόμαστε κλιματισμό εδώ, να λειτουργεί ο κλιματισμό χωρί να τον έχουμε ανάγκη. Δεν χρειαζόμαστε σήμερα κλιματισμό. Όλα έχουν σχεδιαστεί προτινάμε να έχουμε φθηνή ενέργεια. Αλλά πληρώνουμε αυτή τη στιγμή το κόστο για όσε λαθασμένε αποφάσει πήραμε πριν από χρόνια. Έχετε λοιπόν δίκιο και θα σας υποστηρίξουμε πολύ σε ό,τι αφορά ε, τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτικής πολιτική τη κοινή αλευτική πολιτική, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα σέβονται το περιβάλλον και είναι πραγματικά θεμελιώδη σημασία να το επιτύχουμε αυτό μέσα στα επόμενα χρόνια ε, μας αναφέρετε ε, τρεις, ε, τρεις μεγάλους τομείς ε, πολιτικής. Αλλά ποιε θα είναι οι κύριε, οι βασικέ πρωτοβουλίε τι οποίε θα λάβετε, για παράδειγμα στο πλαίσιο τη ε, πολιτική για τη βιοπικιλότητα. Ποιε ακριβώ πρωτοβουλίε θα λάβετε, τι θα κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πέρα από το να λέει πόσο σημαντική είναι η βιοπικιλότητα. Το ίδιο σε ό,τι αφορά την ε, οικονομική διαχείριση των πόρων. Τι ακριβώ θα κάνουμε. Και μετά αναφερθήκατε στην ποιότητα του αέρα. Ε, θα καλύψετε και την ε, έρευνα που λαμβάνει η χώρα σε ό,τι αφορά τον ε, αέρα εσωτερικών χώρων. Γιατί νομίζω πως υπήρχε μια πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εσεί υποτίθεστε να τη δώσετε μια συνέχεια. Ευχαριστώ, λέω ο πρόεδρος, Κρι Ντέιβι τώρα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μπράντι σε αυτόν τον αγίο της συζήτηση, πρόεδρε. Ευχαριστώ Κρίστη, ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ε, μάλλον σαφή παρουσίαση που έκανε και την έκθεση των προτεραιοτήτων του. Θεωρώ πως είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα εργασιών του. Και ζητήσατε, Επίτροπε, την ε, βοήθειά μας και τη χρειάζεστε και χαίρομαι για το γεγονός ότι ξεκινήσατε την παρουσίασή σας αναφερόμενος στην ε, σημασία της βιοπικιλότητας ε, και εγώ θα αναφερθώ στην εμπειρία που αποκόμισα ε, στην διάσκεψη ΣΥΤΕΣ πριν από δύο εβδομάδες. ΣΥΤΕΣ είναι από τα λίγα φόρα για την βιοπικιλότητα όπου έχουμε διεθνή αν θέλετε και το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διάσκεψης ήταν πολύ κακό και το ένα από τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν ότι δεν είχε κανένας είδους επίδραση η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Ε, και αυτό οφείλεται στους οργανωτικούς λόγους, καθώς ε, τα κράτη-μέλη δαπανούσαν 5-6 ώρες την ημέρα για να οργανωθούν, να συντονιστούν μεταξύ τους, ξεχνώντας ότι υπάρχουν 150 χώρες ακόμα οι οποίες συμμετέχουν εκεί ε, και των οποίων συνεργασία χρειάζεται για να επιλυθούν τα προβλήματα της βιοποικιλότητας. Ένα ακόμα ζήτημα ήταν ότι άργησε τόσο πολύ να καταλήξει στην κοινή της ε, θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε ο, η, ο Ιάπωνας Υπουργός ήταν σε θέση να επισκεφθεί ε, άλλες ε, αντιπροσωπείες άλλες χώρες. Άρα λοιπόν από άποψη διπλωματικής, αν θέλετε, πολιτικής διπλωματίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι να αναμένουμε από εσά, θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί πλέον, πιο ισχυροί ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές μας ικανότητες και τη χρήση άλλων εργαλείων πέρα από την επιστημονική μας υποστήριξη, δηλαδή χρηματοδοτική και ούτω καθεξής θα έπρεπε να κάνουμε κάτι. Θα το πάσει, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε τον Επίτροπο που βρίσκεται σήμερα εδώ για να συζητήσει μαζί μας. Μία εβδομάδα πριν από το Πάσχα βρίσκα στο Ελσίνκι μαζί με τον Επίτροπο Τατζάν και ανακοινώσατε τρεις μείζονες συμφωνίες σε ό,τι αφορά τον κανονισμό ΡΙΤΣ ε, προκειμένου να ξεφύγουμε λίγο από το αντιέξοδο στο οποίο είχαμε οδηγηθεί τον τελευταίο καιρό. Ήταν πολύ θετικό αυτό, αλλά Όπω γνωρίζετε πολύ καλά, τα μεγάλα προβλήματα προκύπτουν πάντοτε στι λεπτομέρειε. Και υπάρχουν κάποιε λεπτομέρειε οι οποίε κατά την δική μα άποψη δεν είναι πολύ ε, θετικέ. Δηλαδή, ε, αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία που ανακοινώσατε δεν καλύπτει τα όσα έχει ζητήσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, καταρχήν, ε, η ουσίες ε, που προκαλούν ιδιαίτερα υψηλή ανησυχία. Υπάρχουν δηλαδή 500 ε, περίπου ουσίες οι οποίες πληρούν αυτή την περιγραφή και εσείς αναφερθήκατε σε 106 ουσίες ε, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες οι οποίες θα προσθεθούν στον λόγο κατάλογο των ουσιών δηλαδή που προκαλούν ιδιαίτερα υψηλή ανησυχία. Αλλά τότε θα έχουμε περίπου 135 ουσίες συνολικά. Άρα 350 ουσίες θα αρχίζουν να μην περιλαμβάνονται, να λείπουν από αυτόν τον κατάλογο. Ερωτώ λοιπόν, εάν συνεχίζουμε αυτού του ρυθμού προσθήκη, αν θέλετε, ουσιών στον κατάλογο, θα χρειαστούμε 10 ακόμα χρόνια, ούτω ώστε όλε αυτέ οι ουσίε ε, που προκαλούν ιδιαίτερα υψηλή ε, ανησυχία ε, περιληφθούν. Οπότε. Η ερώτησή μου είναι γιατί χρειαζόμαστε ένα τόσο μεγάλο χρόνο διάγραμμα, δηλαδή τόσο μεγάλο βάθος χρόνου. Τέλο χρόνου, λέει ο πρόεδρο, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο πολύ πολύ σύντομα να μα πει, γιατί αλλιώ δεν έχουμε χρόνο. Ναι, είναι δύσκολο βέβαια αυτό, γιατί είναι πολύ πολύπλοκα τα ερωτήματα που μου θέσατε. Κύριε Ζέμπερ, για το νερό, που είπατε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο επίπεδο. Ναι, θα πρέπει να το προσπαθήσουμε αυτό και ποτέ δεν είχαμε αντίθετη πρόθεση για τα θέματα επικοινωνία. Σωστά το είπατε. Χτε συζητήσαμε το τι θα πρέπει να γίνει με τον Κάρελ. Όταν έκανε τις διαπραγματεύσεις για τη σλοβενική προσχώρηση, είχαμε δημοσιεύσει ένα άρθρο αν κάποιος θα ήθελε να συνδράμει. Και δύο μόνο πλευρές είχαμε που ανταποκρίθηκαν από το περιβάλλον και από τη γεωργία, από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι λοιπόν ε, καλό αυτό και καταδεικνύει ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει γόνιμο έδαφος επίσης. Ε, μια δραστηριότητα η οποία προάγεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας μου για τον καθαρισμό και την απολύμανση των ναρκοπαιδίων. Είναι καλή αυτή η πρωτοβουλία. Κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα κάνουν, αναλαμβάνουν τέτοιε δράσει ε, επιτόπου, όχι μόνο από κεντρικό επίπεδο διακυβέρνηση. Προ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε για του γενετικά τραποποιημένου οργανισμού. Έχετε δίκιο είναι ένα ερώτημα το οποίο ακούω συχνά. Ξέρετε. Ότι αυτό είναι απόκειτα στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ε, όλοι οι αρμόδιοι για θέματα γάμματα α, όμικρον μετέβησαν ε, στη σχετική συνάντηση αλλά είναι αρκετά αδύναμη η θέση μας σήμερα. Έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά και πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στα θέματα αυτά, τα οποία συνδέονται με τους ε, γενετικά τραποποιημένους οργανισμούς και με το περιβάλλον και ξέρω ότι θα πρέπει να συμμετάσχω ενεργά σε τέτοιες συζητήσεις στους κόλπους της Επιτροπής. Άρα θα πρέπει να αναπτύξουμε εκ νέου τις δραστηριότητές μας, όχι στο ίδιο επίπεδο όπως πριν, αυτό είναι σαφές, αλλά χρειαζόμαστε σαφώς κάποιους οι οποίοι θα εξετάσουν και αυτή την πτυχή για το περιβάλλον. Η κυρία Μακέβαν. Νομίζω ότι ένα από τα, μία από τις συγκεκριμένες ε, απαντήσεις που μπορώ να σας δώσω, αν διαβάσετε και την ομιλία μου για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, θα δείτε και θα δείτε μάλιστα ότι δεν είναι η θέση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έχω συζητήσει φυσικά και με τον συνάδελφο Κάλλας ε, και συμφωνεί και αυτός της, με τη λογική αυτή που προασπίζω. Είναι απλή η λογική. Αν υπάρχουν αγρότες, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Πεθρός, δάση και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Υπάρχει λοιπόν Υπάρχουν οι αγρότες στις εκμεταλλεύσεις αυτές, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, για την οποία πληρώνονται. Αλλά αν πραγματικά μας απασχολούν η βιοπικιλότητα, τα ύδατα, το έδαφος, θα πρέπει να θεωρήσουμε τις υπηρεσίες τους ως κοινοφελείς υπηρεσίες και θα πρέπει να τις αποζημιώνουμε για αυτές. γιατί ακούγονται εκεί κάποιες φωνές κατά της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τις αντικρουόμενες αυτές απόψεις προκειμένου να καταλήξουμε σε μια κοινή αγροτική και περιβαλλοντική πολιτική, όπως ανέφερα στην ομιλία μου. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτό θα αποδώσει καρπούς. Ας περιμένουμε να δούμε τη στρατηγική για την βιοπικιλότητα, γιατί θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα από τα πλέον δύσκολα έγγραφα τα οποία θα, πρέπει, να προετοιμάσουμε για φέτος, αλλά δεν θέλουμε να, να τηρήσουμε μεροληπτική στάση σε ό,τι αφορά την βιοπικιλία. Πρόσφατα εκφώνησα και μια άλλη ομιλία, την οποία μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μου. Αλλά στον τομέα αυτό θα ήθελα να περιμένω λίγο ακόμα, να ακούσω και άλλες ε, απόψεις προτού αποφανθώ για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικού χώρου βρισκόμαστε σε πρώιμη φάση, αν σωστά κατάλαβα. Είσαστε κι εσείς ε, επιτόπου και είδατε Πώ δεν πρέπει να εφαρμόσουμε τη στρατηγική τη Λισαβόνας. Είναι το καλύτερο μάθημα που πήραμε αυτό. Καταρχάς, ως κοινότητα δεν είμαστε μέλος του ΣΥΤΕΣ. Είναι μυστική η ψηφοφορία, δεν ξέρουμε και ούτε καν πόσοι ψήφισαν. Ελπίζουμε όμως να ψηφίσουν όπως συμφωνήσαμε. Επίση, είναι σημαντικό να αλλάξει η κατάσταση και να μιλήσουμε με μία φωνή. Κατά δεύτερον, όντως χάσαμε όλο το χρόνο που χρειαζόμασταν για διπλωματικές δράσεις για τις δραστηριότητε μας. Από πλευράς της Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλουμε τις προτάσεις. θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι προτάσεις αυτές από την προηγούμενη Επιτροπή. Ξέρετε ότι, ότι αποφασίσαμε με την κυρία Ταμανέκη σε μία ημέρα. Σε μία ημέρα καταλήξαμε σε απόφαση γιατί θέλαμε να υπάρχει κάποιος χρόνος για την καλή μεταφορά των όσων συμφωνήσαμε. Αλλά τα κράτη-μέλη χρειάστηκαν δύο-τρία κορεπέρ προτού τελικά καταλήξουν. Εμείς ευχαρίστως να πάμε στη διεθνή συνάντηση με την κοινή μας θέση. Αλλά εντωμεταξύ οι άλλοι εταίροι, η Ιαπωνία, η Κίνα κάνουν λόμπι ασκούσαν έντονες πιέσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό λοιπόν δεν μας ικανοποιεί. Και επίσης έγιναν κάποιες καλές προτάσεις από κράτη-μέλη, τις οποίες με τις οποίες δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, με τις οποίες εγώ προσωπικά θα συμφωνούσα πάρα αυτά αν ε, αποφάσιζα μόνος μου, αλλά δεν είχαμε σχετική εντολή. Μάθαμε πάντως θεωρώ ότι δεν είναι σωστός τρόπος αυτός να προχωρήσουμε θα μπορούσαμε να έχουμε καταλήξει σε σωστέ συμφωνίες στο ιστορικό τη Ένωση, αλλά αποτύχαμε σε διεθνές επίπεδο και τελικά αποτύχαμε μια τρύπα στο νερό. Για το συνδυασμό των ξένων μέσων συμφωνώ, θα ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικά. Αλλά θεωρώ ότι αυτό μεταφέρει μεγάλο τμήμα της ευθύνης στην ΕΚΑΔ, στην Επιτροπή για την αλληλεία. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή και σίγουρα θα το συζητήσω με τον συνάδελφο. Με τη συνάδελφο νομίζω όμως ότι η κυρία Δαμανάκη αντιλαμβάνεται πολύ σωστά τη σοβαρότητα του θέματος. Για το ρίτς τέλος. Ξέρετε, θα μπορούσε κανείς να πει με ευκολία ότι τον δυσαρεστεί ή τον ευχαριστεί. Αλλά μετά από τρία χρόνια ακινησίας, αν κάποιος ε, βγει και πει ότι είναι ικανοποιημένο, αυτό τι να σας πω, με προβληματίζει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να περάσω στην εφαρμογή του REACH και θεωρώ προσωπικά ότι τα όσα συμφωνήσαμε με τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη είναι ωφέλιμα για το περιβάλλον. Να επαναλάβω ορισμένα εξ αυτών, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι τι περιλαμβάνεται στην Συμφωνία REACH. Καταρχάς, συμφωνήθηκε να μην υπάρξει παράταση της πρώτης προθεσμίας του 2010. Κατά δεύτερον, το παράρτημα υπαριθμό 13 συμφωνήθηκε ότι όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να εξεταστούν σε ό,τι αφορά την ε, ταυτοποίηση VTB, GPT αυτό θα αποτελέσει μια νέα απέτηση για τη βιομηχανία. Αποφασίσαμε λοιπόν να περιλάβουμε μεταβατικά μέτρα προκειμένου να δώσουμε στον κλάδο το χρόνο που χρειαζόταν για να τα εφαρμόσει. Και επίσης αποφασίσαμε το συντομότερο δυνατό να περάσουμε σε καθεστώς επιτροπολογίας. Βρίσκεται λοιπόν αυτό υπό εξετασή στην Επιτροπή. Και όταν λέμε το συντομότερο δυνατόν εννοούμε πάρα αυτά στην συγκεκριμένη περίπτωση. Κάτι το οποίο επί δυόμιση χρόνια βρισκόταν σε ακινησία. Συμφωνώ επίσης μαζί σας ότι έχουμε πολύ πιο πολλά. Ίσως να είναι 500 οι ουσίες αυτές, χίλιες, δεν ξέρω. Αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχει συμφωνία για τον αριθμό αυτό. Υπάρχουν σαφώς πολύ πιο πολλές. Πολύ πιο πολλά στοιχεία από αυτά που προτείνουμε. Σε τρία χρόνια, ως τώρα, είχαμε 29 στην, το κατάλογο των υποψηφίων. Και τώρα προσθέτουμε 43 έτος, το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, την, αν, την ανώτατη ποσότητα που μπορεί να απορροφηθεί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ΕΚΑ θα πρέπει να απασχολήσει πιο πολύ προσωπικό, αλλά... Μην θεωρείτε ότι αν δημιουργηθεί μια καινούργια υπηρεσία από το 2007 θα καταστεί και λειτουργική και να σας πω ότι χρειάζονται τουλάχιστον τρία χρόνια όσο του καταστεί μερικώς λειτουργική μια τέτοια επιχείρηση γιατί δύο σχετικές ε, υπηρεσίες που έχω παρακολουθήσει ακόμα δεν είναι πλήρως λειτουργικές. Δική μου φιλοδοξία φυσικά είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία και να συμφωνήσουμε επί ενός οδικού χάρτη Το σχέδιο υποκατάστασης, το οποίο είναι το τελευταίο στοιχείο. Συμφωνήσαμε ότι αυτό ισχύει και, και για τον σωστό α, έλεγχο και για τον σωστό οικονομικό και κοινωνικό έλεγχο. Αλλά έτσι όπως έχει η νομοθεσία σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί μεροληπτική. Άρα θα μπορούσαμε να περιμένουμε καταρχάς ίσως ένα χρόνο προκειμένου να δοθεί σαφής νομική ερμηνεία ή η άλλη δυνατότητα να ξεκινήσουμε την εφαρμογή και ξεκινήσαμε, για να ξεκινήσει μάλιστα με τρόπο για το σωστό έλεγχο η υποκατάσταση, ενώ στην άλλη περίπτωση να γίνει προσωμείωση της υποκατάστασης. Λίγο πολύ το ίδιο, αλλά με διαφορετικό όνομα. Θα δημοσιευτεί ένα σχετικό έγγραφο στην επίσημη εφημερίδα. Θα μεταφραστεί δηλαδή και στις 27 γλώσσες, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν πρόσβαση στη δική τους γλώσσα. Σας ε, ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά ήταν απαραίτητα αυτά. είναι ενδιαφέροντα τα όσα. Θα ακούσουμε και σχετικά στο Ελσίνκι, καθώς θα τα πούμε και αύριο λοιπόν. Αντές περίλου, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα δάση. Έχουμε γνωρίσει διάφορα πρόγραμματα δράση και την πράσινη βίβλο, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε 27 πολιτικέ στην Ευρώπη αλλά ούτε καν δύο, μία για το Βορρά, μία για τον Νότο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στην Κομισιόν υπάρχει ε, άποψη για μια ενιαία ολοκληρωμένη πολιτική αναφορικά με τα ευρωπαϊκά δάση, θεωρώντας τα ευρωπαϊκά δάση ως μια ε, ενότητα και ε, αν προτίθεστε να αναπτύξετε μια τέτοια πολιτική θεωρώντας ότι τα, θα υπά, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει τα δάση ανά την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριε Σπέτερλε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας σήμερα εδώ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν αναφέρεστε σε μια πιο ευρεία πολιτική. Και αναφερθήκατε ε, και εσείς όπως και άλλος επιτρέπω σε αυτή την αλλαγή στο παράδειγμα, δηλαδή στην προσέγγιση, τη λογική που ακολουθούμε και θα ήθελα να ακούσω από εσά ε, τι ακριβώς ε, επιθυμεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να επιτύχουμε περισσότερο πρόοδο, περισσότερη πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ εσάς και του Τρούπερινγκ να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Θέσατε πολύ φιλόδοξους στόχους στον εαυτό σα σε ό,τι αφορά την ε, ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ε, και κάνουμε ταυτόχρονα όμως λόγο για την κατασκευή νέων μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν με βάση το λιγνίτη. Πώς ακριβώς λοιπόν θα επιτύχετε πρόοδο. Επίσης μιλήσατε και για κάποια νέα προϊόντα Καθώς ε, λοιπόν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τον προηγούμενο επίτροπο και ήσασταν επίτροπο επιστήμη. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, ποιες είναι οι αλλαγές που θα δούμε. Μιλάμε δηλαδή για όραμα εδώ, άρα ε, πώς θα επιτύχουμε στον χώρο, για παράδειγμα, του ηλεκτρισμού ένα ε, καινούριο επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά το νέο Ινστιτούτο, πραγματικά μπορούμε να ελπίζουμε πως θα υπάρχει κάτι εδώ, θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα έδειμο που θα διευκολύνει τα νέα προϊόντα. Κύριος Δέβης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ε, ζητήματα θα ήθελα να θέσω. Ε, σε ό,τι αφορά την οδηγία και την εκάψη των αποβλήτων. Έλαβα μόλι τώρα μία απάντηση από τη δική, απάντηση από τη δική σας πλευρά και πραγματικά ήταν πολύ θετική σε ό,τι αφορά τη μείωση δηλαδή των εκπομπών γιατί έχει ε, μειωθεί, έχουν μειωθεί οι σχετικέ διακοπέ κατά 200 φορέ. Δηλαδή, ουσιαστικά ε, η εκπομπή διοξενών έχει ουσιαστικά ελαχιστοποιηθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εφαρμογή τη οδηγία εδώ τη νομοθεσία γίνεται με το σωστό τρόπο, είναι αποτελεσματική. Επιστρέφοντα τώρα στο REACH αφού αναφέρθηκε σε αυτό και ο πρόεδρο, Πραγματικά είχαμε ένα σωρό προβλήματα, σχέδια δράση, τα οποία τελικά δεν είδαμε πού ε, οδήγησαν που δώσαμε προτεραιότητα σε αυτές τις διαδράσει. Θα ε, μπορούσαμε ενδεχομένω να το θέσουμε αυτό και την αρμόδια υπηρεσία για τα γιατί ε, βλέπουμε έρθρα, άρθρα στι εφημερίδε όπω αυτό στην ε, Δανία, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις Ζενόλη, η οποία, οποία ακόμα χρησιμοποιείται στα παιδικά μπερό και πρόκειται να απαγορευτεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή, υπάρχουν ε, κάποιοι φόβοι οι οποίοι προκύπτουν στη μία στην άλλη χώρα, αλλά χρειαζόμαστε μια λογική προσέγγιση, γιατί βλέπουμε πως ε, εδώ δεν έχουμε επιτύχει την πρόοδο που θα επιθυμούσαμε σε ό,τι αφορά κάποιους μακροπρόθεσμους ε, στόχους που έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Ο Σάντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πριν από λίγα λεπτά μας είπατε ότι χρειαζόμαστε μια καθαρή βιομηχανία και δεν χρειαζόμαστε μόνο καθαρές ή μάλλον χρειαζόμαστε καθαρές τεχνολογίες και όχι τεχνολογίες που καλούνται εκ των υστέρων να καθαρίσουν τρόπο την άτηση υπάρχουσες. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά θα ήθελα να σας ε, αναφερθώ σε μια συγκεκριμένα τεχνολογία στον χώρο των, των εξορίξεων και εγώ τόσο όσο και ο συνάδελφος ε, Τρεμόπουλος είχαμε απαιτηθεί σε εσάς ε, μια ερώτηση, μια και μας δώσατε μια πολύ τυπική απάντηση. Υπάρχουν και άλλες πολιτικές ομάδες όπως οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλιστές και ε, κάποιοι ευρωβουλευτές από το ΕΛΚ που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το ζήτημα. Ε, είχατε ήδη αναφερθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης θέας σε αυτό το ζήτημα ε, και το ερώτημά μου τώρα είναι το εξή. Σε δύο εβδομάδες το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί στο Στρασβούργο και θα υπάρξει μια σχετική συζήτηση. Υποστηρίζετε εσείς την απαγόρευση της εν λόγω τεχνολογίας, δηλαδή τη χρηστοσάνατος μέσα στην ε, εξωτερική βιομηχανία, στη θετική τεχνολογία. Χρειαζόμαστε εδώ μια επανάσταση σε όρους λογικής την οποία ακολουθούμε. Σας υποστηρίζω στις προσπάθειές σας να απαγορεύσετε από τους συναδέλφους σας να αποστέλουν απλώς και μόνο τυπικές απαντήσεις. Ε, παίξτε δηλαδή εδώ έναν ε, βασικό τέτοιο ρόλο. Ο κ. Ασένης έχει το λόγο. Thank you very much. And, ε, Ευχαριστώ. Χαιρόμεθα που βρίσκεστε ανάμεσά μας και που συζητήσατε το θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Μιλάμε για τις κλιματικές αλλαγές και όλοι προσπαθούμε να βρούμε μια νέα όθηση μετά από την αποτυχία της Κοπεχάγης. Το ζήτημα που μας απασχολεί είναι η αποψήλωση, κάτι το οποίο οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, επίσης έχουμε φασίσει την ε, οικονομική ενίσχυση των ε, δασών αυτών. Η Κομισιόν όμως έκανε μια πρόταση σχετικά με την παράνομη ξυλία, αλλά δεν την απαγορεύει. Και έτσι αν τα ξυλία εισάγεται από περιοχές όπου εφαρμόζεται η παράνομη λοτομία και δεν μπορούν να υπάρξουν οι κατάλληλοι έλεγχοι, αυτά, τα, αυτή η ξυλία θα ε, πολίτες τους ε, Ευρωπαίους καταναλωτές. Λέγεται επίσης ότι δύσκολα θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη μια απαγόρευση και θα πρέπει να ελέγχεται όλες οι ποσότητες ε, ξυλίας ε, που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας ερωτώ, το κόστος της ε, απαγόρευσης είναι τόσο υψηλό ώστε να επιτρέπουμε την ύπαρξη μιας νομοθεσίας η οποία περιλαμβάνει τόσα πολλά κενά. Καλχάινς Φλόρενς. Καλώς ήρθατε εδώ. Κύριε Επίτροπε, έχουν υποθεί καλά λόγια για εσά. Συμφωνώ και εγώ με αυτά. Ε, εμένα με ανησυχεί ξανά και ξανά η εφαρμογή ε, κανόνων που έχουμε αποπαθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μας είπατε ότι θα ε, ε, λάβετε εδώ πιο αυστηρά μέτρα, θα κάνετε πιο αυστηρά βήματα. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι ακριβώ εννοείται για όλα αυτά τα οποία επιθυμούμε να κάνουμε, τα Triple και οτιδήποτε άλλο. Εκεί δηλαδή είχαμε ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το ότι είχαμε μια πολύ καλή ιδέα η οποία όμω εφαρμόστηκε με πολύ πολύ άσχημο τρόπο. Και εδώ δεν μιλάω για τα νέα κρατημέλη, μιλάω για τα παλαιά κρατημέλη. Κυρία ε, Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, η Κοπεχάγη αποτέλεσε αποτυχία. Φυσικά δεν είστε υπεύθυνο για θέματα κλίματος, ε, αλλά μας απαντάτε σε θέματα που μπορούν την πράσινη ανάπτυξη. Τώρα, σε ό,τι φορά την Κοπεχάγη, το πακέτο για, μιλούσε για έναν έλεγχο στα σύνορα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προτιμούν να μην ε, δεσμευτούν σε μια νομοθεσία αναφορικά με το κλίμα, αλλά θέλουν να, έχουν, να εφαρμόσουν μια, μια βολονταριστική πολιτική καινοτόμα. Λοιπόν, περιμένουμε τις ε, προτάσεις του Πρόεδρου της Επιτροπής κ. Μπαρόζο σχετικά με τις συνέπειες της Κοπενχάγης. Λοιπόν, ποια είναι η θέση σας ε, αναφορικά με την ιδέα ενός μηχανικού, ενός μηχανισμού που θα ε, περιλαμβάνει ελέγχου στα σύνορα και το, μια που μιλάτε για πράσινη ανάπτυξη, ποια είναι η οικοκαινοτομία, η οικοανάπτυξη και πώς προβλέπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ, γιατί σήμερα στο πλαίσιο της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διανύουμε, βλέπουμε τις ΗΠΑ και την Ασιατική Ήπειρο να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και η Ευρώπη να ε, καθυστερεί. Πώς λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε μετά από την αποτυχία της Κοπενχάγης, ε, τι θα να κάνουμε για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά ταυτόχρονα να υλοποιήσουμε και να αναπτύσσουμε μια πραγματική βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Κυρία Γκουτιέρες, ευχαριστώ πολύ. Μου άρεσε η παρουσία σας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομία και την απασχόληση. Να κάνω δύο ερωτήσεις πρώτα απ' όλα. Με ενδιαφέρει το ζήτημα της βιοποικιλότητας, αλλά με ανησυχεί το ότι δεν ε, μιλάμε για το ότι η βιοπικιλότητα ε, συνδέεται με την υγειοργία και τα υδατά. Ξέρουμε ότι τα πτηνά πίνουν νερό. Αλλά βλέπουμε ότι και αυτή η κατάσταση επηρεάζει και την αναπαραγωγή των πτηνών αλλά και των ζώων. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σημαντική πτυχή την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεύτερον, μου δόθηκε εντύπωση ότι η οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν λάμβανε υπόψη την ε, ιστορική κληρονομιά μας. Ίσως διότι οι ενδιαφερόμενοι είναι βιολόγοι. Αλλά έχω δύο σημαντικά ζητήματα να πω εδώ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση που σέβεται την έννοια της ιστορικής κληρονομιάς, γιατί στην οδηγία την οποία εξετάσαμε χθε για την απαγόρευση συγκεκριμένων προϊόντων και τη χρήση του ε, στα, ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές συσκευέ, δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την ε, ιστορική κληρονομιά. Μιλάμε για την αισθητική των ε, κτηρίων. Θα χρειαστεί να κλείσουμε κάποια μουσεία και να μην μπορέσουμε να ανακοινήσουμε κάποια κτίρια για λόγους ασυμπατότητας. Νομίζω ότι διακόπτει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα επίσης να ακούσω ότι και διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε κ. ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που παρουσίασε τα σχέδιά του για τα επόμενα χρόνια σας και χαιρόμαστε που αναφέρεστε στην εξοικονόμηση των πόρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως να διευρυνθεί η ατζέντα γιατί διαβάζονται στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι περιοριζόμαστε στην χρήση της ενέργειας. Θα θέλαμε λοιπόν να διευρυνθεί αυτή η ατζέντα, να μιλήσουμε και για τη χρήση των γεών, τη χρήση των υλικών, των ε, μετάλλων, γιατί χρειάζεται σχετική ατζέντα και για το θέμα αυτό. Τι εννοούμε όμως με την ε, αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων, γιατί εξακολουθεί να επικρατεί η αύξηση των της χρήσης ε, γεών και υδάτων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Και επίσης, ε, στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε με πάρα πολλούς επιτρόπους. Θα πρέπει να συνεργαστείτε με πολλές επιτρόπους, με πολλές ομάδες εντός της Επιτροπής. Θα είναι δύσκολο το έργο αυτό. Και ως Κοινοβούλιο θα σας υποστηρίξουμε γιατί δεν πρόκειται να είναι εύκολη η συνεργασία αυτή. Μία συγκεκριμένη ερώτηση. Σήμερα, στην παρούσα φάση, μιλάς, μιλούμε για τη βιωσιμότητα της χρήσης της βιοενέργειας. Πόσο συγκεκριμένα εργάζεστε στην παρούσα φάση, προκειμένου οι σχετικέ πολιτικές της Ένωσης να αποδώσουν καρπούς και πώς θα συνεργαστείτε με τον κύριο Ιτενγκερ, με την κυρία Χέριγκαρτ, για να διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει η βιωσιμότητα αυτή και σε ό,τι αφορά την έμεση αλλαγή της χρήσης των γεών. Ευχαριστώ. Η κυρία Φαμπρέντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω και να πω ότι έχετε την απόλυτη και αμέριστη συμπαράστασή μας σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών. Να σας ρωτήσω για τα δύο απόβλητα. Κάτι πολύ συγκεκριμένο στις ε, συζητήσεις που γίνονται στις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Με απογοητεύει κάπως το γεγονός ότι δεν έχετε αποφανθεί ακόμα, δεν έχετε αποστείλει ένα σαφές μήνυμα το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το οποίο θα λάβει την υποστήριξη και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Τρεις ε, προεδρίες έχουν ταχθεί υπέρ σαφών οδηγιών για τα βιοαπόβλητα. Αλλά είναι αντικρουόμενα τα μηνύματα τα οποία ακούμε από τη δική σας υπηρεσία και ο Γενικός Γραμματέας Day δήλωσε ότι δεν είναι υπέρ ξεχωριστής ε, οδηγίας για τα βιοαπόβλητα και θα πρέπει ότι, είναι υπέρ της προσαρμογής ε, κάποιων άρθρων για τις οδηγίες για τα απόβλητα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ανεπαρκές. Είμαι βέβαιη ότι και εσείς συνειδητοποιείτε τη μεγάλη σημασία των δύο αποβλήτων σε ό,τι αφορά την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων αυτών. Και θεωρώ ότι αυτό για να μπορέσει να περάσει χρειάζεται μια ξεχωριστή οδηγία η οποία θα αναφέρεται όχι μόνο στην ανακύκλωση, αλλά θα προβλέπει και σαφή κριτήρια ποιότητας, κριτήρια συλλογής των αποβλήτων αυτών. Δηλαδή, να θέσει ένα σαφές πλαίσιο. Μία απλή ερώτηση λοιπόν. Είσαστε υπέρ μια τέτοια ε, ξεχωριστή οδηγία και σκοπεύετε να υποβάλλετε μια τέτοια πρόταση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και όπω βλέπετε, Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, Τώρα ακούσατε πιο πολλές ερωτήσεις για να τις απαντήσετε όλες μαζί. Είναι σημαντικό να θέσουν τα ερωτήματα τους οι συνάδελφοι. Ο κ. Τρομόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις για δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα αφορά το θόρυβο μια και η οδηγία του 2002 απαιτεί από τα κράτη-μέλη να κάνουν χαρτογράφηση για τα επίπεδα του θορύβου. Απαιτεί κάθε πενταετία η Επιτροπή να δημοσιεύει συνοπτική έκθεση σχετικά με τα δεδομένα των κρατών που περιλαμβάνονται στους χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης. Απαιτεί επίσης η οδηγία το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουλίου του 2009 η Επιτροπή να έχει υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ε, οδηγίας με εκτίμηση της ανάγκης για παραπέρα κοινοτικέ δράσεις σχετικά με τον περιβάλλοντα θόρυβο και να προτείνει στρατηγικές. Η έκθεση του Συμβούλου αναμένεται τέλη Μαΐου. Μπορείτε, κύριε Επίτροπε, να διαβεβαιώσετε την Επιτροπή μας ότι προτίθεστε να υποβάλλετε την πρόταση για αναθεώρηση ε, με δεσμευτικά όρια ελάχιστης προστασίας ή ανώτατα όρια έκθεσης προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει μέτρα αντιμετώπισης μεγάλων πηγών χορύπανσης όπως ε, τα αεροπλάνα, το δικό, το κατασκευαστικό δίκτυο και ο κλάδος. Επίσης, ε, κύριε Πίτροπε, δηλώσατε στις 18 Μαρτίου ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμορφωθούν γρήγορα με τα κοινοτικά πρότυπα ποιότητας του αέρα και να μειώσουν τις εκπομπές τους. Στις γραπτές απαντήσεις ε, στις 13 Ιανουαρίου είχατε δηλώσει ότι θα προχωρήσετε σε αναθεώρηση της οδηγίας των ανώτατων εθνικών ορίων εκπομπής εν ώψη των φιλόδοξων στόχων του 2020. Επειδή οι αέριοι ρήποι είναι δολοφονικοί, προκαλούν τουλάχιστον 370.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο. Thank you. Thank you Γιατί... δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας η... Ε, Not more right than the others, please. Two words, Mr. Przepraszam bardzo, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Panie Komisarzu, ja mam pytanie dotyczące sieci Natura 2000, o której Pan tylko... Έχω μία ερώτηση σχετικά με το δίκτυο Natura 2000. Αναφερθήκατε, απλώς το θίξατε ακροθήγως θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ιδρύσαμε αυτό το δίκτυο προκειμένου να λάβουμε υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και την αηφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων που ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το δίκτυο Natura 2000 έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κρατημένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις το δίκτυο αυτό ομιλικά περιέπλεξε ή κατέστησε αδύνατη την οικονομική ανάπτυξη κάποιων ε, κοινοτήτων. Ε, παραδείγματος χάρη δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε δρόμους, ε, υπονόμους κλπ. Γι' αυτό έχω δύο ερωτήσεις. Ποιες, ποιοι είναι οι στόχοι σας, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας ε, σχετικά με την διαχείριση αυτού του συστήματος Natura 2000 του δικτύου. Και δεύτερη ερώτηση πώς ε, θα έχει η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον λογοδίκτυο. Ευχαριστώ. Μακίνες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας έκανε. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα ήθελα να ακούσω περισσότερα είναι ότι δεν γίνεται τιμολόγηση προϊόντων τροφίμων, για παράδειγμα. Δεν περιλαμβάνεται το συνολικό τους κόστος. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό, γιατί σε ό,τι αφορά την γεωργική πολιτική αποφασίσαμε ότι η αγορά έχει αποτύχει. Αλλά εσείς δεν θα πρέπει να ομολογήσετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα, δεν υπάρχει ένα σύστημα όπου η αγορά αποτυπώνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής των προϊόντων αυτών και θα ήθελα πιο πολλά τέτοια στοιχεία και σε ό,τι αφορά και το ΕΚΑ. Να ακούσουμε τι πιστεύετε για το REACH. Λέτε ότι η υπηρεσία αυτή λειτουργεί και ότι πρόκειται για ένα επαναστατικό βήμα από πλευρά ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για τα χημικά. Είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε από, να διδαχτούμε από άλλους, αλλά τουλάχιστον ίσως μπορέσουμε να διδάξουμε άλλους στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Σιώκενσεν. Thank you and, and also thank... Σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την εξαιρετική του παρουσίαση και τις πολύ λεπτομερείς απαντήσεις που μας έδωσε. Μία ερώτηση για την ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Είπατε ότι θέλετε να διασφαλίσετε ένα ισότιμο επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. Πολύ με απασχολεί όμω ότι αυτό θα αποτελέσει τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, γιατί στη χώρα μου οι πολιτικοί μας συζητάνε κατά πόσο θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις προθεσμίες Λένε δηλαδή αιρετή πολιτική στη χώρα μου ότι εφόσον δεν θα τηρήσουν άλλε χώρε την προθεσμία, γιατί να την τηρήσουμε εμεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό ο σωστό τρόπο για την εφαρμογή. Πώ θέλετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον, Πιστεύετε ότι έχουμε ακόμα ε, ευκαιρία να ανταπεξέλθουμε και να τηρήσουμε την προθεσμία του 2015 σε ό,τι αφορά την πολιτική και τα ύδατα. Thank you, Christa ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της βιωσιμότητας ε, ως ζήτημα προτεραιότητας, αλλά πρόκειται εδώ για διατομεακές, για οριζόντιες αρμοδιότητες ε, και πράγματι η βιωσιμότητα αποτελεί συχνά εξισορρότησα ε, μεταξύ διαφορετικών παραγόντων. αναφερθήκατε στα βιοκτώνα και στο γεγονό ότι θα έχουμε μια κοινή νομοθεσία, κοινέ ρυθμίσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πράγματι εδώ αυστηρότερα όρια, αλλά προβλέπονται και ορισμένε εξαιρέσει. Για κάποια δηλαδή προϊόντα τα οποία μπαίνουν σε, σε ένα κατάλογο για υποκατάσταση, αλλά ενδεχομένω θα χρειαστούμε τέτοια προϊόντα. Άρα λοιπόν πώ θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το, το ενδιαφέρον τη οικονομία για τέτοιου είδου προϊόντα. Πρόκειται λοιπόν για ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες ε, αξιώσεις σε ό,τι αφορά την υγεία και από εκεί και μετά υπάρχει και, ε, υπάρχουν και κατάλληλες σε ό,τι αφορά το κόστος. Θα αναθεωρηθεί το σχετικό κόστος. Ε, και μετά η σχετική υπηρεσία θα αναλάβει τις σχετικές αρμοδιότητες, θα, θα λάβει και τους απαραίτητους πόρους ώστε να μπορέσει να ασχοληθεί και με αυτό το ζήτημα των βιοκτών. Κάτι τέτοιο θα ήταν, πολύ, ε, θα ήταν κάτι το πολύ θετικό, θα ήταν μια μεγάλη πρόοδος δηλαδή να έχουμε έτσι μια τέτοια πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Ευχαριστώ Λεπρόεδρος, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Εξετίμησα ιδιαίτερα την παρουσίασή σας, ε, ιδίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ε, απόδοσης και αποτελεσματικότητας των πόρων. Αυτό θα μπορούσαμε να το με μια πρόταση πολύ σύντομη ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι, όπως είναι περιορισμένη και η, δυνατότητα της γης ε, να μεταβολίζει τα απορρίμματά μας. Αυτές είναι οι δύο βασικές εκφράσεις που εγώ ονομάζω ένα reset, μια διόρθωση, μια ε, αναδιάρθρωση της κοινωνίας μας. Αυτή οι δύο περιορισμοί λοιπόν θα πρέπει να μας ε, οδηγήσουν σε μια αλλαγή πολιτισμού, μια πολιτισμική αλλαγή. Δεν πρόκειται για ζήτημα περιβάλλοντος πλέον, ε, αλλά η πολιτική συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει από τη δική μας Επιτροπή και από την συνεργασία μας. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα πιο εξειδικευμένα, όπως η προστασία του εδάφους, σας ζητάω να εξετάσετε το ζήτημα αυτό και να κάνετε μια συστημική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της περιβαλλοντικής αλλαγής, της κλιματικής αλλαγής, εννοώ και θα πρέπει να δοθεί η ασφάλεια και η διασφάλιση αυτού του κοινού αγαθού το οποίο θα προκύψει από την διαχείριση. Πάντως θα αποδεχθώ την ανοιχτή θύρα και τη διαθεσιμότητά σας για συνεργασία. Ευχαριστώ. Νομίζω πως είχαμε εδώ μια μεγάλη γκάμα ερωτήσεων. Α, όχι, έχουμε και άλλους ομιλητές. Συγγνώμη. Έχουμε και άλλους λοιπόν. Κύριος ε, Θεόδωρος Τιλακάτης έχει το Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για την, ε, πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ε, μιλήσατε εκτεταμένα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική χρήση των πόρων και υπάρχει μια ακόμα πιο θεμελιώδης αρχή στην νομοθεσία μας, δηλαδή αυτή του ο ρηπαίνων πληρώνει. Δηλαδή αυτό προορίζεται και προβλέπεται και στην σχετική νομοθεσία για τις επιδοτήσεις ε, σε ό,τι αφορά τον άνθρακα. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή εφαρμόσουμε την ε, αρχή του ο Ριπένον πληρώνεται, όχι πληρώνει. Θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε αυτή την επιδότηση των ορεικτών καυσίμων. Ευχαριστούμε, κυρία Εστρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να πω ότι η στρατηγική 2020 είναι πολύ χρήσιμη και σημαντική <clears throat> για την περιβαλλοντική πολιτική, διότι πρέπει να αλλάξουμε οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης στην Ευρώπη. Και για τον λόγο αυτό η στρατηγική θα πρέπει να είναι το δυνατόν φιλόδοξη. Έχουμε ανάγκη από την αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας μας για να διασφαλίσουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Έχουμε ανάγκη από μια ενεργειακή πολιτική η οποία θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στην ενεργειακή απόδοση, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή μας πολιτική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσατε βραχυπρόθεσμα να προτείνετε προκειμένου να αυξηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άρα να καταστήσουμε πιο ανεξάρτητη και αυτόνομη την Ευρώπη από τον εφοδιασμό της από τρίτες χώρες. Κύριο Σόνικ έχει το λόγο. Δεν θέλετε να μιλήσετε, εντάξει. Ευχαριστούμε. Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Ε, η οδηγία για τα εδάφη ε, γεννήθηκε και απεβίωσε άμεσα τώρα ε, η συνάδελφος κυρία Δαμανάκη που είναι υπεύθυνη για την θαλάσσια πολιτική και την αλία ε, της ε, ετέθη μια ερώτηση σχετικά με την συνεκτική με τη συνέπεια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα συνεργαστείτε μαζί της και τι είδους συντονισμό προβλέπετε, αφενός από την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που προβλέπει κάποιους ενιαίους χώρους θαλάσσιους και την δική πολιτική, την ε, στρατική για το θαλάσσιους ε, περιοχές και τις παράκτιες περιοχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, εντυπωσιάστηκα ομολογουμένως από τον φιλόδοξο τόνο της ομιλίας της αλλά και από το ιδιαίτερα ρεαλιστικό πρόγραμμά σας. Και αυτό το πρόγραμμα σίγουρα θα οδηγήσει την Ευρώπη σε ένα πράσινο μέλλον. Όλοι στην Ευρώπη σας υποστηρίζουμε. Αλλά επίσης υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι γνωρίζουν πώς τα προγράμματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν. Θα ήθελα να θίξω το ζήτημα του κόστους. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό, διότι το κόστος είναι υψηλό. Πάντως, θα πρέπει να πείτε σε κάποιες βιομηχανίες ότι υπάρχουν καλύτερες μέθοδοι και καλύτερες τεχνικές που θα, θα τους βοηθήσουν στο να πάψουν να χρησιμοποιούν ε, κιάνιο. Thank you, Mr. Chairman. Ε, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, κυρία Μορκενάιτε, σας ευχαριστώ, Επιτροπέ, για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας και προφανώς ήταν δύσκολο να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, αλλά να σας ρωτήσω κάτι για την μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Ακούμε να ανακύπτουν τακτικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μεγάλων προγραμμάτων, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Και τα πιο πολλά προβλήματα προέρχονται από την έλλειψη ε, διαφάνειας και την έλλειψη ε, αμεροληψίας και η κοινωνία θέλει πιο διαφανείς κανόνες για την εφαρμογή των ε, μελλοντικών αυτών μελετών αντικτύπου για το περιβάλλον. Τι πιστεύετε, είναι δυνατόν να υπάρξει ένα μέσο προκειμένου να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους περιβαλλοντικούς ε, με περιβαλλοντικές μελέτες αντικτύπου. Η κυρία Βάσκερ δεν θέλει το λόγο πλέον. Ωραία, ολοκληρώσαμε λοιπόν. Και τώρα... Είπα εξ αρχής ότι είναι σημαντικό να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Είναι αδύνατον φυσικά να απαντήσετε στα πάντα. Μπορείτε να απαντήσετε και γραπτά, οπότε επίτροπε επιλέξτε εσείς ε, την ερώτηση που θεωρείτε πιο σημαντική, τις ερωτήσεις που θεωρείτε πιο σημαντικές. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, δεν αρκούν. Βλέπω πόσο έντονα έχετε επεξεργαστεί το έγγραφο αυτό με τόσα χρώματα. Νομίζω ότι έχετε επισέλθει σε λεπτομέρειες τις οποίες δεν μπορείτε να παρουσιάσετε, τις οποίες θα λάβουμε όμως από τον Έχετε το λόγο. <coughs> Uh, αυτό είναι και ο μοναδικό τρόπο για να μπορέσω να προχωρήσω, διότι έχω πέντε σελίδε ερωτήσεων, όχι απαντήσεων. Πες το, θα προσπαθήσω να τι διατρέξω εντάχει τώρα για την προστασία των δασών και την ενημέρωση. Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, κάτι το οποίο έμαθα και πολύ γρήγορα είναι φυσικά κρίνω ότι τα δάση έχουν τεράστια σημασία και θα πρέπει να τα δημιουργήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχουν σημαντικές ε, αντιστάσεις που προέρχονται από κράτη-μέλη σε επίπεδο ε, συζητήσεων ε, και επικουρικότητας ε, τώρα σε ό,τι φορά την συνεργασία με τον κύριο Έρτεγκερ. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Μπορέσαμε να συνεργαστούμε και οι δύο ε, δείχνουμε ανοιχτό πνεύμα και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη. Όταν συζητάτε ε, από εθνική σκοπιά σε αυτό το μείγμα ενέργειας ε, και το οποίο αποφασίζεται από τα κράτη-μέλη, είναι κάτι το οποίο, παραλαμβάνω, βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Και ο λόγος είναι απλός. Οι δομές ε, στα κράτη-μέλη διαφέρουν σημαντικά. Και φυσικά δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις πολιτικές τους, αλλά Θεωρώ ότι η στρατηγική της ενέργειας και των τεχνολογιών είναι πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν η στρατηγική γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα ζήτημα επιπλέον, διότι γνωρίζω πολύ καλά τι βρίσκεται πίσω από την ερώτηση και ξέρετε ότι και εγώ ήμουν σαφής συζητώντας το ζήτημα στην χώρα μου είναι ότι κάθε χώρα όταν λαμβάνει απόφαση σχετικά με το ενεργειακό μείγμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο. Και αυτές είναι σοβαρές δεσμεύσεις και <clears throat> που συνδέονται με, το θέμα όχι μόνο του 2020 αλλά και τη θετική του 2050. Σήμερα μιλάμε για μια μείωση της κατα κατά 20-30% αλλά μιλάμε μέχρι το 2020 αλλά μιλάμε για μείωση 80% μέχρι το 2050 όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κύριε Ντέιβις εδώ υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα ενώπιον μπροστά μου πάνω στο ζήτημα αυτό και στο πιο σημαντικό ζήτημα είναι ότι η Κομισιόν έχει ξεκινήσει μελέτες ε, για την για να λάβει υπόψη τα τελευταία επιτεύγματα <clears throat> στην αλλά και τις τελευταίες ε, επιστημονικές έρευνες ε, που έχουν γίνει. κύριος Έντελ πήσε και ερώτηση κύριο Παναγιώτου για το ωκεάνιο. Δεν μπορώ να σας ε, δώσω μια πολιτική δέσμευση, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα εργαστούμε πολύ σοβαρά για την εξέταση του ζητήματος, διότι θεωρώ είναι πολύ σημαντικό όλες οι αποφάσεις μας να στηρίζονται σε σαφείς απόψεις. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει κάπου, αλλά θα δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, η αποδάσωση δέουσα επιμέλεια ή όχι. Αυτό δεν ρωτήσατε. Α, όχι, απαγόρευση. Απαγόρευση ή δέουσα επιμέλεια. Να σας πω για ποιο λόγο η απαγόρευση θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει κανένα, καμία σχέση με τη φιλοδοξία εξάλλου. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι η επιμέλεια είναι μια πιο συστηματική προσέγγιση χωρίς να χρειάζεται να ελέγχουμε κάθε φορτίο. και θα οδηγήσει σε υψηλό κόστος η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την παράνομη ε, υλοτομία σε, τρίτα, σε τρίτο κράτος θα είναι σχεδόν αδύνατον και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να κρίνει εάν έχει παραδιαστεί νομοθεσία τρίτης χώρας, κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνο με την παράδοσή μας. Τώρα, η Δέουσευ επιμέλεια με ρωτάτε αν θα επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε όταν κάναμε την αξιολόγηση αντικτύπου και η απαγόρευση ήταν κάτι που μας ε, απασχόλησε. Αλλά όπως σας είπα, αποφασίσαμε τη δόση επιμέλεια, διότι θεωρούμε ότι η εφαρμογή της απαγόρευσης ε, ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί. Ο κ. Φλόρενς αναφέρθηκε στο ζήτημα της εφαρμογής να πω ότι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά δουλεύουμε και προχωράμε βήμα προς βήμα και μας απασχολεί ιδιαίτερα η κυρία Γκροστέτ για την Κοπενχάγη. Ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σοβαρό είναι εντάξει, η Κοπενχάγη ήταν μια χρεοκοπία γνωστό σε όλους. Και πρόσφατα έγινε μια ανακοίνωση που αναφέρει ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής. Μην υποτιμάτε το γεγονός ότι οι υπόλοιποι δεν εργάζονται πάνω στο ζήτημα αυτό της ε, κλιματικής αλλαγής. Εγώ ασχολήθηκα με το θέμα της έρευνας και της ε, ανάπτυξης και να σας πω ότι οι Αμερικανοί, Κινέζοι, οι Άπωνες συμμετέχουν σημαντικά για, στο ζήτημα αυτό της ε, κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να το έχουμε λοιπόν αυτό κατά νου. Κριστίνα Κουτιέρες. Βιοπικιλότητα, γεωργία, συμφωνώ απόλυτα. Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας <clears throat> αυτό το ζήτημα που αναφέρεται ρητά. Στην οδηγία τώρα το αρχή κληρονομιά που δεν λαμβάνεται υπόψη το καταγράφω και το κατανοούμε πως είναι σημαντικό. Κύριε Σπάς, ε, ε, αποτελεσματικότητα των πόρων, συζητώντας το ζήτημα αυτό, συχνά καταλήγαμε ε, με στο θέμα της ε, ενεργειακής απόδοσης. Φυσικά η αποτελεσματικότητα των ε, πόρων είναι κάτι το ευρύτερο από την ενεργειακή απόδοση τώρα. Ενεργειακές πολιτικές και αηφορία και εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη την Ουγγαρία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση λεπτομερώς, αλλά θεωρώ ότι η αηφορία των πολιτικών είναι ζωτική σημασίας Και για μένα ο μοναδικός τρόπος ε, για να λυθεί το ζήτημα είναι κάθε ζήτημα να το εξετάζουμε σε βάθος, ε, εξετάζουμε, βρίσκουμε, κάνουμε αναλύσεις ε, αντικτύπου, αξιολόγηση αντικτύπου. Διότι διαφορετικά τα πράγματα γίνονται με τρόπο συναισθηματικό και δεν είναι πάντα αποτελεσματικά. Τώρα για τα δύο απόβλητα. Νομίζω ότι δεν τίθεται το θέμα αν είμαι εγώ υπέρ ή όχι. Το θέμα είναι τι υποδεικνύουν τι καταδεικνύουν οι μελέτες αντικτύπου που έχουμε κάνει ως τώρα και επίσης, όπως είπατε, δεν μπορώ να γνωρίσω και την, ε, τις αντίθετες φωνές που ακούγονται στην Επιτροπή που καλούν για επικουρικότητα. Αυτά είναι τα γεγονότα, αυτά έτσι έχει η πραγματικότητα. Η δική μου ανησυχία σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για τα βιοαπόβλητα είναι ότι αφενός υπάρχουν τα στοιχεία που καταδεικνύουν οι μελέτες δεκτύπου, που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, που λένε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για νέα νομοθεσία. Και αυτό είναι το βασικό που θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την τρέχουσα νομοθεσία και να προσθέσουμε κάποια στοιχεία. Όταν κοιτάμε την ε, οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα δεν εφαρμόζεται. Αν είχε εφαρμοστεί θα λαμβάνονταν υπόψη τα στοιχεία αυτά για τα παράνομα ναρκοπαίδια. Και πάλι, αν εφαρμόζονταν σωστά η νομοθεσία, πολλά στοιχεία θα ρυθμίζονταν. Να προσέχουμε λοιπόν όταν ζητούμε νέα νομοθεσία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για το περιβάλλον και αυτό θα πρέπει να κοιτάμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Όχι με υπερβολική ρύθμιση. Και θεωρώ ότι στην περίπτωση αυτή θα τύχανε αυτό της υποστήριξη κάποιων κρατών μελών, γιατί έτσι θα αναβάλλονταν, αναφέρεται θα λάμβαναν καινούργιε προθεσμίες για την εφαρμογή τη ήδη φυστάμενης νομοθεσία. Λέει ο Πρόεδρος, βλέπω ότι καλύψαμε τις 2,5 από τις πέντε σελίδες, θα πρέπει να κλείσουμε όμως, να προτείνω να κλείσουμε εδώ τα δύο απόβλητα. Σα ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις που μας δώσατε και νομίζω ότι οι υπόλοιποι θα λάβουν τις απαντήσεις τους κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας για την δέσμευσή σας. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε και θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και στο μέλλον. Να έρχεστε στην Επιτροπή μας όποτε θέλετε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. 26 Απριλίου η επόμενη συνάντηση πέρα της συναντήσεις.